colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω να αρχίσουμε, γιατί έχουμε ήδη κάποια καθυστέρηση. Δεν θα σας παρακαλέσω να καθίσετε στις θέσεις σας και να περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν θα να σας ενημερώσω ότι προτιθέμεθα το σημείο 7 η γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ήτρε για την καινοτομία θα το συζητήσουμε αύριο και σήμερα ανταυτού να συζητήσουμε το θέμα 10. Εάν δεν διαφωνεί κανένας θα αλλάξουμε τη σειρά αυτή και ελπίζω να μπορεί να εγκριθεί η ημερησία διάταξη με αυτές τις μικρές αλλαγές και να περάσουμε στο σημείο 2 της ημερησίας διάταξης που είναι η έγκριση των πρακτικών της περασμένης μας συνεδρίασης στις 22 Φεβρουαρίου. Θα να προτείνω, εάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν διαφωνήσει κανένας, θα θεωρήσουμε εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 της μέρης διάταξης, ανακοινώσεις Προέδρου. Και θα ήθελα καταρχήν να σας ενημερώσω ότι μέσω της γραπτής διαδικασίας που ξεκίνησε μετά την περασμένη μας συνεδρίαση, οι συντονιστές αποφάσισαν να προτείνουν την εξή χορήγηση μια έκθεση και μια γνωμοδότηση. Η έκθεση για την πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ελλανδία έχει χορηγηθεί στο ΕΛΚ και θα ήθελα ο συντονιστής να ορίσει κάποια από τα μέλη του ΕΛΚ γι' αυτό. Να πω το, το όνομα. Σαν Κέλλη είναι. Σας το λέω αυτό. Το δεύτερο είναι, είναι γνωμοδότηση για την απασχόληση στο μέλλον κοινωνικών υπηρεσιών. Οι σοσιαλδημοκράτες θα ορίσουν κάποιον. Δεν έχουμε όνομα ακόμα. Σας παρακαλώ λοιπόν να ενημερώσετε τη γραμματεία το γρηγορότερο δυνατόν σχετικά. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω αφορά τον τρόπο με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να οργανώσει τις αντιδράσεις του για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Υπήρξε μια συνεδρίαση που οργανώθηκε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, στην οποία συγκάλεσε 7 ή 8 προέδρους ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών, που θεωρούνται ίσως πιο σχετικές προς το σχέδιο αυτό του 2020. Είχαμε ένα δείπνο εργασία κατά τη διάρκεια του οποίου εκφράστηκαν πρώτα σχόλια για την στρατηγική αυτή. Τα κύρια θέματα αφορούσαν μάλλον τις διαδικασίες και όχι την ουσία. Και όσον αφορά τις διαδικασίες, η γενική η ιδέα ήταν ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στην πραγματική συζήτηση του 2020 γιατί το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των στρατηγικών είναι πάρα πολύ στενοποιημένο. Οι συζητήσεις θα αρχίσουν στο Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και θέλουν να υιοθετήσουν το έγγραφο αυτό κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορφής του Ιουνίου. Και μεταξύ Κομισιόν εργάζεται πάνω στις κατευθύνσεις γραμμές ο ρόλο του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ περιορισμένο στο έγγραφο που έχει υποβάλει η Κομισιόν, που πιστεύουμε ότι δεν είναι ευθυγραμμισμένο με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθούν σημαντικέ προσπάθειες από πλευρά του Κοινοβουλίου, αυτή είναι το δράση δική μου άποψη, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αυξήσουμε τον ρόλο μας, να τον ευθυγραμμίσουμε δηλαδή με τη συνθήκη, γιατί εκπροσωπούμε τους πολίτες της Ευρώπης και μιλάμε εξ ονόματος των πολιτών της Ευρώπης στη συζήτηση για τη στρατηγική αυτή. Μερικοί από τους συναδέλφους θα από τον Πρόεδρο να, να βάλει τη διαδικασία αυτή και να υιοθετηθεί η στρατηγική μετά το καλοκαίρι. Άλλοι από εμά που είμαστε πιο ρεαλιστές λέμε ότι έχει εκκινηθεί όλη η διαδικασία και υπάρχει και ένα αίσθημα κατεπήγοντος. Ε, και γι' αυτό οι πιθανότητες να μην γίνει δεκτό από τη διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου είναι πολύ μικρές. Πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μα. Συζητήσαμε επίση πώ θα οργανωθούμε και εμεί και το Κοινοβούλιο για τη ζήτηση για το 2020. Υπήρχαν διαφορετικέ απόψει. Μια επιτροπή ad hoc, μια διευθύνουσα επιτροπή και είδε επίσης η διάσκεψη των Προέδρων να είναι το βήμα στο οποίο θα οργανωθεί αυτή η συζήτηση. Αυτό ήμουν ανοιχτό κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασία που σας προενέφερα. Την επόμενη μέρα η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε όσον αφορά το θέμα αυτό και ζητήθηκε από τη διάσκεψη των ε, Προέδρων των ε, Κοινοβουλευτικών Επιτροπών να οργανώσει τις εργασίες μας για το 2020 και από ό,τι κατάλαβα η διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα προτείνει μια, ένα χρονοδιάγραμμα για την οργάνωση των εργασιών του Κοινοβουλίου για το 2020. Αυτή είναι η κατάσταση που ήθελα να σας παρουσιάσω. αυτά είχα να σας πω. Ο Λάμπερ Φανιστερό ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Με κάποιους συνδυασμούς, Πρόεδρε, έχω να πω, είναι σαφές ότι είναι ασαφή τα πράγματα. Είναι περίεργο ότι αυτή τη στιγμή που ξεκινάμε ε, με ένα νέο συμβούλιο, με μια νέα επιτροπή, αδεχόμαστε αυτούς τους περιορισμούς. Αν θυμάμαι σωστά, θέλαμε να έχουμε κάποια θέση, να τοποθετηθούμε δηλαδή. Και εμείς σαν Επιτροπή, όλα αυτά λοιπόν δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Και αν υπάρχουν πραγματικά καινοτομίε στην προετοιμασία, γιατί να μην αφιερώσει δύο μέρες το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, με μια νέα διαδικασία. Ε, τώρα εντάξει, έχουμε την διάσκεψη των Προέδρων των ε, Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Αλλά όλα αυτά είναι εκ των άλλων προς τα κάτω, έτσι δεν είναι. Γιατί λοιπόν να μην εφεύρουμε μια νέα διαδικασία. Να είμαστε πιο ευέλικτοι. Να έχουμε δύο μέρες προετοιμασίας και μετά ένα ψήφισμα. Δεν έχουμε τις δυνατότητε αυτές και αναρωτιέμαι. Πιστεύετε ότι το ΕΕ 2020 θα προσφέρει περισσότερη συνοχή και δέσμευση στο μέλλον μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης ε, αν δεν έχουμε προετοιμαστεί καλύτερα. Όχι, το ίδιο θα έχουμε. Λοιπόν, θα έχουμε το ίδιο και μετά θα έχουμε νομικές ε, προτάσεις, προτάσεις νομοσχεδίων και θα τις μπλοκάρουμε εμείς. Λοιπόν, καλύτερα να έχουμε δύο μέρε χωρί συγκεκριμένη ημερησία διάταξη να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Αυτό εδώ πέρα που προτείνεται δεν είναι καλά ισορροπημένο μεταξύ αυτό που θέλουμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Πρώτα, σας ευχαριστώ Λαμπέρ. Κάποιο άνθρωπος θέλει να πάρει το λόγο. Θα επανέλθουμε βέβαια στο 13 αύριο στο θέμα αυτό. Εκεί έχουμε την συζήτηση ε, της έκθεσης Κόρτες Λάστρα για τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην επίδευση των στόχων της Λισαβόνας. Αλλά εγώ ζήτησα από την ε, διάσκεψη των Πρόεδρων Κοινοβουλικών Επιτροπών να αλλάξει τον, τον τίτλο Δηλαδή να συμπεριλάβουμε όχι μόνο τις αντιδράσεις ε, για την Λισαβόνα, αλλά και μέσα στα πλαίσια του 2020. Και περιμένουμε από αυτού την απόφαση της διάσης των Προέδρων, που ελπίζω θα είναι θετική. Και έτσι ίσως μπορέσουμε πραγματικά το Μάη να έχουμε μία συζήτηση που θα ξεκινήσουμε εμείς μέσα στα πλαίσια της Συνόδου. Και πριν από μερικές εβδομάδες έστειλα και μία επιστολή στη Διάστηση των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ε, όσον αφορά την ανάγκη να υπάρχει αυτή η συζήτηση για την Ευρώπη του 2020. Για Γιάννη το λόγο. Με συγχωρείτε που ήρθα με καθυστέρηση, αλλά ένα αντίστοιχο σχόλιο είναι, διαβάζοντας πολύ προσεκτικά την τελευταία εκδοχή της στρατηγικής του 2020, λέγεται ξεκάθαρα ότι η στρατηγική αυτή ανήκει στα χέρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και λέει, ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι να προετοιμάσει την, την νομοθεσία για τη στρατηγική του 2020, αλλά η ιδιοκτησία, αν θέλετε, της διαδικασίας αυτής παραμένει στα χέρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι καλό να το ξέρουμε. Αυτό υπάρχει στο κείμενο, όπως σας είπα. Πρόεδρος. Καλά, εντάξει, νομίζω ότι θα μπορούμε να επανέλθουμε στη συζήτηση αυτή στο σημείο 13, όπως σας είπα, και ακόμα αργότερα. Δεν μπορούμε τώρα να δεχθούμε, βέβαια, κάποιες από τις προσεγγίσεις όσον αφορά ιδίως το ρόλο του Κοινοβουλίου στην ε, στρατηγική του 2020. Υπάρχει νομοθετική εργασία, υπάρχει και το θέμα της προώθησης ε, του 2020 όταν χρειαζόμαστε συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ωραία, λοιπόν. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια αυτή τη στιγμή και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4. Η πρώτη έκθεση του Μιχάλη Τρεμόπουλου. Πού είναι ο Μιχάλης? Α, εδώ, ναι. Δεν είστε ποτέ εδώ μαζί μας. Αλλά έτσι σας βλέπω τουλάχιστον. Ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη συζήτηση για το σχέδιο έκθεσης. Θα υπάρχει και προθυμία για τις τροπολογίες. Ήθελα να δώσω το λόγο στον Μιχάλη όμως, θα μας κάνει μια Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ε, γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 2005 την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την ε, Διαφάνεια, το ETI. Και ακολούθησε η δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου το 2006. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης. Η παροχή δημόσιας πληροφόρησης σχετικά με τους δικαιούχους των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πρωτοβουλίας αυτής. Όσον αφορά τη δημοσίευση των δικαιούχων των διαρθρωτικών ταμείων, και του Ταμείου Συνοχής, η υποχρέωση αυτή καθορίζεται από τον κανονισμό της Επιτροπής που ρυθμίζει τους κανόνες για τα διαρθρωτικά ταμεία. Το άρθρο 7.2 Δέλτα απαιτεί τη δημοσίευση πληροφοριών τριών κατηγοριών. Πρώτα τον κατάλογο των δικαιούχων, μετά τα ονόματα των επιχειρήσεων και τρίτον το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και των διαχειριστικών αρχών όσον αφορά την ερμηνεία αυτών των ελάχιστων απαιτήσεων της ε, Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια. Αντικατοπτρίζουν διαφορές τόσο στις διοικητικές ικανότητες καθώς και στις πολιτιστικές και διοικητικές παραδόσεις και νοοτροπίες. Για να το πούμε κομψά. Αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις κατέστησαν δυνατές από το σχετικά χαλαρό νομικό πλαίσιο που φυλάσσει την υποχρέωση της δημοσίευσης στοιχείων σχετικά με τους δικαιούχους. Η Επιτροπή περιορίζει το ρόλο της αρχικά στο να προτείνει ένα κοινό ενδεικτικό πρότυπο για τη δημοσίευση των στοιχείων και αφετέρου να παράσχει στο κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες μέσω του ιστοτόπου της ε, περιφερειακής πολιτικής, το DG Regio, με συνδέσμου για ηλεκτρονικέ διευθύνσει των κρατών μελών όπου δημοσιεύονται τα απαιτούμενα δεδομένα σχετικά με του δικαιούχου των Ευρωπαϊκών Ταμείων Περιφερειακή ανάπτυξη και του Ταμείου συνοχή. Υπό το καθεστώς κοινή διαχείριση των διαθροτικών ταμείων, αυτέ ε, οι συνδέσεις και το περιεχόμενό του, είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και βασίζονται σε πληροφορίε που παρέχονται από τι διαχειριστικέ αρχέ η μεταβλητότητα στην παρουσίαση και στις συνθήκες πρόσβασης στα δεδομένα δεν επιτρέπουν την πλήρη σύγκριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, προτείνω στο σχέδιο έκθεσης η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτές τις βάσεις δεδομένων των κρατών μελών και την αναζήτησή τους πλήρως συμβατές, ώστε να διευκολυνθεί μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση των στοιχείων που παρουσιάζονται, διατηρώντας παράλληλα το τοπικό ενδιαφέρον. Από την άποψη αυτή θα μπορούσε να εξεταστεί η χρήση δύο γλωσσών, της τοπικής ή των τοπικών γλωσσών και στα αγγλικά. Παρόλο που κανένα μέλος δεν δημοσιεύει λιγότερα δεδομένα από αυτά που ορίζουν οι ελάχιστες απαιτήσει, αν και ορισμένα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας δεν συμμορφώνονται πλήρως, Παρ' όλα αυτά λοιπόν ορισμένα κράτη-μέλη επιλέγουν τη δημοσιοποίηση πρόσθετων πληροφοριών, όπως οι στόχοι των σχεδίων, οι ομάδες στόχοι στην περίπτωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Ταμείων, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απέτηση που ορίζεται στο ισχύο νομικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, το προτινόμενο σχέδιο έκθεσης τονίζει ότι η χρησιμότητα των στοιχείων που προβλέπονται για τις ανάγκες των δικαιούχων πρέπει να βελτιωθούν τόσο όσο αφορά το περιεχόμενο όσο και την παρουσίαση. Καλή λοιπόν την Επιτροπή να καθορίσει μια πιο λεπτομερή και κανονιστική μορφή προσδιορίζοντας τη δομή, τη μορφή και το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται. Η συνολική ποιότητα του συστήματος γνωστοποίησης θα μπορούσε να ενισχυθεί παραπέρα αν οι γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη μοιράζονται από κοινού τους κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές. Απευθύνει επίσης το σχέδιο έκκληση για πρόσθετες βασικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά τη δημοσίευση των καταλόγων των δικαιούχων, ε, όπως η τοποθεσία και τα συνολικά στοιχεία επικοινωνίας, τις περιλήψεις των εγκεκριμένων σχεδίων, είδη στήριξη καθώς και περιγραφή των εταίρων του σχεδίου. Η διεθνής διαφάνεια έχει επικρίνει την αδιαφάνεια των κονδυλίων αυτών, καθώς έχει προσδιοριστεί επίσης ως κίνδυνος διαφθοράς και εμπόδιο για τον προσδιορισμό ευθυνών. Ως αντίλογος σε αυτή την άποψη, προβλήθηκε ότι η οικονομική στόχη που προκαλεί η αδιαφανής εκταμίευση και ένα αντίστοιχο σύστημα αναφοράς είναι λιγότερο επιβαρυντική από τις διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από τη συστηματική γνωστοποίηση των δικαιούχων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποκάλυψη των στοιχείων για τα κονδύλια όμως επιτρέπει την συμμετοχή του κοινού σε μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο που δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της δημοκρατίας. Η προετοιμασία της πολιτικής συνοχής για την εποχή μετά το 2013 θα πρέπει να πάρει υπόψη στο το γεγονός ότι η πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσει της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια θα μπορούσε να εξασφαλιστεί καλύτερα μέσω της ισχυροποίησης των κανονισμών και των κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Στα πλαίσια του αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης, η διάχυση των πληροφοριών αποτελεί βασικό στοιχείο της ορθής διαχείρισης και ελέγχου. Βοηθά στην πρόληψη προβλημάτων που ανακύπτουν και την προώθηση της συμμόρφωσης. Το άρθρο 69 του Γενικού Κανονισμού για τα Διαρθωτικά Ταμεία αναφέρει ότι το κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των ταμείων. Ο εκτελεστικός κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία κοινού δικτύου υπευθύνων επικοινωνίας με αρμοδιότητα σε επίπεδο διαχειριστικής αρχής. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το δίκτυο Inform για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε, η συνοχή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται επίσης μέσω μιας συμβουλευτικής δομής της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων. Ενισχύει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά μεταξύ των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων και τονώνει την εθνική συνεργασία στην προώθηση της στήριξης της διαρθρωτικής χρηματοδότησης. Μέσα από τον καθορισμό των δικτύων αυτών και τη συλλογική τους πίεσης, η Επιτροπή υιοθετεί μια προσέγγιση προς την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας προώθησης για τη διαφάνεια και όχι την επιβολή του κανονισμού σχετικά με τις διαχειριστικές αρχές, ενώ είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να εγγυώνται την ακρίβεια των δημοσιευμένων στοιχείων. Στο σχέδιο έκθεσης καλούμε την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια θα πρέπει να τεχθεί σε εφαρμογή σε επιχειρησιακούς όρους στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και σχεδίων επικοινωνίας τους. Επιπλέον, τονίζω τη σημασία της ορθής και έγκαιρης παροχής πληροφοριών από τα κράτη-μέλη ως αποτρεπτικό μέτρο στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου και συνεπώς η ανάγκη να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια και των οικονομικών ελέγχων και των ελεγκτικών μηχανισμών. Επαναλαμβάνω τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξέφραζε, εξέφρασε στο ψήφισμά του στις 19 Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διαφάνεια στα δημοσιονομικά θέματα ότι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πρέπει επίσης να καλύπτει τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Προτείνω επίσης την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ανακτήσεις και τις αποσύρσεις σύμφωνα με την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στο σύνολό τους. Επιπλέον, το σχέδιο έκθεσης καλεί την Επιτροπή να κρατήσει μια πιο σκληρή γραμμή για την επικοινωνία και τις απαιτήσει πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων και της τακτικής κατονομάζω και διαπομπεύω και τη χρήση των δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια πρέπει επίσης να έχει σημαντική επίδραση για τους κανόνες μιας διαφανούς εταιρικής σχέσης στις προς τα άνω και τις προς τα κάτω φάσεις της διαδικασίας προγραμματισμού. Η συνεργασία πρέπει να συμβάλλει στη διαφάνεια, την υπευθυνότητα, την αποτελεσματικότητα και νομιμότητα σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού, της συνοχής και της εφαρμογής. Το σχέδιο έκθεσης ζητεί ως εκ τούτου τα κράτη-μέλη και οι διαχειριστικές αρχές για τη συμμετοχή των εταίρων, περισσότερο σε όλες τις φάσεις σε ένα πρώιμο στάδιο και να τους δώσει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα του έργου με σκοπό να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεών τους η εταιρική σχέση μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων από το γεγονός και μόνο ότι θα επιτρέπεται στις διαχειριστικές αρχές να έχουν πρόσβαση στη γνώση βασισμένη σε κριτήρια γεωγραφικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της στοχοθέτησης των παρεμβάσεων βελτιώνοντας κατά συνέπεια την απορρόφηση των πόρων και την ποιότητα του έργου. Η εταιρική σχέση μπορεί επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση της λογοδοσίας στο μέτρο που η πράξη εταίρων λειτουργεί ως πομπός και πολλαπλασιαστής του προγράμματος ενημέρωσης για τις εκλογικές τους περιφέρειες, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια. Το άρθρο 11 του Γενικού Κανονισμού για τα Διορθωτικά Ταμεία απαιτεί η εταιρική σχέση να καλύψει τα διάφορα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων. Από την εκπόνηση ως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ωστόσο, πέραν του προημίου του κανονισμού, καθώς και του συγκεκριμένου άρθρου σχετικά με την αρχή της εταιρικής σχέσης, υπάρχει πολύ μικρή αναφορά σε εταίρους ή εταιρική σχέση στις ενότητες περί επιχειρήσεων των ρυθμιστικών κειμένων και δεν παρέχονται ακριβείς και επίσημα δεσμευτικές οδηγίες ή καθοδήγηση από την Επιτροπή σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης. Με αυτόν τον τρόπο, η πραγματική ερμηνεία του τρόπου συμμόρφωσης προς το άρθρο 11 επαφίεται στις αρχές των κρατών μελών και κατά συνέπεια η εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης εξαρτάται από τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές. Και κακές συνήθειες θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Δεδομένου ότι ο ρόλο τη Επιτροπή φαίνεται να είναι υπερβολικά παθητικό και περιορίζεται στην παρατήρηση, το σχέδιο έκθεση, ζητά περισσότερε κατευθυντήριε γραμμέ από την Επιτροπή σχετικά με το πώ θα τεθεί η ρήτρα για την εταιρική σχέση στην πράξη, για τα τρέχοντα προγράμματα και για αρκετά δεσμευτικού κανόνε για την εταιρική σχέση στα μελλοντικά κανονιστικά κείμενα. Καλή επίση για την παροχή της καλύτερης στόχευση και πιο τακτικής ενημέρωσης σε οργανισμούς εταίρους, καθώς και για την ενισχυμένη χρήση της τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της εταιρική σχέσης, μεταξύ άλλων δίνοντας την ευκαιρία σε οργανώσεις εταίρους να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις κατάρτισης που διοργανώνονται για τα όργανα παράδοσης. Στο σχέδιο έκθεσης επισημαίνω το γεγονός ότι τα ελάχιστα πρότυπα διαβούλευσης είναι ένα στοιχείο της πρωτοβουλίας αυτής για τη διαφάνεια και ότι έχουν προωθηθεί αυτά τα πρότυπα και εφαρμόζονται από την Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Αν εμεί δικαίω ζητούμε μεγαλύτερη διαφάνεια από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, στη συνέχεια τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει επίσης να είναι διαφανή στον τομέα αυτό. Ωστόσο, παρτερούμε αναεπαρκής εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις της Επιτροπής, σχετικά με τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων και συνεπώς μια έλλειψη διαφάνειας που πρέπει να διορθωθεί. Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Γενικού Κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει ή να απορρίψει μεγάλα σχέδια που υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη αφορά προγράμματα με προπολογισμό πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα του περιβάλλοντος ή 50 εκατομμύρια ευρώ σε άλλους τομείς. Η ανοιχτή δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με αυτά τα μεγάλα έργα πριν από την απόφαση για τη χρηματοδότησή τους αποτελεί κοινή πρακτική μεταξύ διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Παγκόσμια Τράπεζα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια εξαίρεση σε αυτόν τον τομέα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο τα πρότυπα διαφάνειας θα πρέπει να είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κάνω έκκληση για την έγκαιρη δημοσίευση των πληροφοριών σε απευθεία σύνδεση online, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πρόσβασης στο έργο τεκμηρίωσης για τα μεγάλα έργα το συντομότερο δυνατόν, αφού η Επιτροπή λαμβάνει αίτηση για χρηματοδότηση από ένα κράτος μέλος και προτού λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την χρηματοδότηση. Αυτή η ιστοσελίδα της Επιτροπής θα πρέπει να επιτρέπει την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με αυτά τα έργα, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να υποφεληθεί από μια ποικιλία πηγών πληροφόρηση σχετικά με τα σχέδια που υποβλήθηκαν, η οποία θα το επιτρέψει να κάνει πιο καλά ενημερωμένους τους πολίτες και καλύτερες αποφάσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι να συμβάλλουμε με αυτή την έκθεση στην μεγαλύτερη διαφάνεια και την καταξίωση των ευρωπαϊκών οργάνων στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Thank you σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε οκτώ ομιλητές. Θα ήθελα σας παρακαλώ να είσαστε επιθαρχημένοι περισσότερο ε, από κάθε άλλη φορά. Κυρία Βέστβαλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως είπε και ο κ. Στρομόπουλος ήδη, η διαφάνεια είναι η έννοια κλειδί για την πολιτική συνοχή, πράγματι. Οι πόροι της ε, ιδιωτικής πολιτικής είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ε, κεφάλαιο στην, ε, στο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει κανένας άλλος τομέας ευρωπαϊκής πολιτικής που έχει άμεσο, τόσο άμεσο αντίκτυπο στους πολίτε, όπως η πολιτική συνοχή. Εμείς ως υπεύθυνοι δεν μπορούμε να δεχθούμε οι πολίτε να αποκτούν την εντύπωση ότι κανένας δεν ξέρει πού προωθούν τα χρήματα αυτά. Γι' αυτό η διαφάνεια ακριβώς στο τομέα της ε, ε πολιτικής είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς, οι σοσιαλδημοκράτες, θεωρούμε ότι ο εισηγητής κ. Τρεμόπουλος παρουσίασε συνολικά ισορροπημένη πρόταση έκθεσης. Οι σοσιαλδημοκράτες ξέρουν ότι οι πληροφορίες για τους παραλήπτες των πληρωμών στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ διαφορετικές και ότι η διαφάνεια ε, ε, ποικίλει από χώρα σε χώρα ταυτόχρονα. η τράπεζα δεδομένων που διαθέτουν τα κράτη-μέλη δεν είναι πάντα πλήρη, πλήρης. Μια ενιαία μορφή αυτών των δεδομένων θα ήταν λοιπόν σημαντική για να πετύχουμε τη διαφάνεια. Πράγματι θα ήταν χρήσιμο εάν οι πληροφορίες δεν μεθύδονται μόνο στην εκάστοτε γλώσσα της χώρας, αλλά τουλάχιστον και στα αγγλικά. Και αυτό θα συνέβαλε στην διαφάνεια. Όσον αφορά όμως το άρθρο 12, το λεγόμενο naming and shaming, εμείς διαφωνούμε με τον εισηγητή. Εγώ είμαι παιδαγωγός α, και στο παιδαγωγικό τομέα δεν εργαζόμαστε πια με την αρχή αυτή της ντροπή γιατί αυτό αντιστρέφεται στο αντίθετό του. Αυτή η παιδαγωγική αρχή δεν οδηγεί πια από ό,τι μάθαμε στον στόχο της. Βέβαια είναι δικαιολογημένη η επιθυμία για μεγαλύτερη διαφάνεια. Την υποστηρίζουμε, αλλά δεν θα πρέπει να οδηγήσει να έχουμε καταλήξει σε ένα κυνήγι μαγισσών. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή, αυτό το σύστημα της κατονομασίας και του νοδισμού, του naming and shaming. Γενικά, οι σοσιαλδημοκράτες εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση της έκθεσης είναι γενικά ισορροπημένη και πάρα πολύ χρήσιμη. Με μονομένε προτάσεις τροπολογίας θα υποβάλουμε προσεχώς. Ευχαριστώ very much. The next speaker is mm-hmm. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον συνάδελφο για την κατάρτιση της ε, έκθεσης αυτής και νομίζω ότι ότι θα πρέπει να επαυξήσουμε την ε, διαφάνεια σε αυτόν τον ε, τομέα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μην θυσιάσουμε την αποδοτικότητα στο βωμό της διαφάνειας. Νομίζω ότι ορισμένες ε, προτάσεις φέρουν ιδιαίτερο βάρος ως προς την εφαρμογή τους και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η περιφερειακή πολιτική στη δική μου επικράτεια στη Γαλλία και θα ήθελα να πω ότι για τις τοπικές αρχές ε, ο φόρτος, ο διοικητικός φόρτος είναι πολύ μεγάλος και η εικόνα που απορρέει ε, δεν συνάδει με την εικόνα της ε, περιφερειακής πολιτικής. Νομίζω ότι θα αναθέταμε έναν επιπρόσθετο φόρτο και θα θέταμε σε δυσκολία αυτή την πολιτική στην καθημερινή της εφαρμογή. Δεν έχουμε ε, χρόνο πολύ. Θα μιλήσω και μαζί σας ε, διμερώς, αλλά θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία. Όταν ζητάτε στο άρθρο 5, στο σημείο 5 πέρα από των ελάχιστων απαιτήσεων να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με τοποθεσία, στοιχεία επικοινωνίας, περιλήψεις. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Ε, επίσης, τα κράτη-μέλη στα πλαίσια του ελέγχου θα πρέπει να δίνουν σαφείς πληροφορίες σε μια συγκεκριμένη προθεσμία. Αυτό θα επιβαρύνει το ολοπλαίσιο κατά της αποδοτικότητας. Νομίζω ότι ορισμένα στοιχεία είναι υπερβολικά σε σχέση με το σημερινό προϋπάρχον πλαίσιο. Κυρίλοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί όπως είπατε έχουμε προβλήματα χρόνου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τρεμόπουλο και το θέμα είναι θέμα εξισορρόπησης μεταξύ διαφάνειας, διαφάνειας χωρίς να επιβαρύνουμε με έναν επιπρόσθετο φόρτο το όλο πλαίσιο. Νομίζω ότι ο τρόπος, με τον τρόπο της απλούστευσης μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την εξισορρόπηση και δέχομαι ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή διότι όλη η διαδικασία είναι ανοιχτή, μπορεί να τύχει καλύτερες διαχείρισης, θα, υπάρχουν, ε, θα υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και παρατυπίες. Και όπως είπανε και άλλοι συνάδελφοι, θα πρέπει να είναι η πολιτική αυτή συνοχής πιο ορατή θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί του γεγονότος ότι ιδιαίτερα για τις νέες χώρες, για τα νέα κράτη-μέλη, οι πληροφορίες είναι αναγκαίες ως προς την αδειοδότηση προγραμμάτων και η δυνατότητα απορρόφησης των αντιστοίχων χωρών πολλές φορές είναι δύσκολη. Όσο αυτή η πληροφόρηση φτάνει στους τελικούς δικαιούχους, τόσο το καλύτερο θα έχουμε μία συνεκτική πολιτική. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ίσως, μάλλον αναφέρεται, αλλά όχι με τον τρόπο που θα επιθυμούσα ίσως εγώ, Αναφέρεται η εφαρμογή ε, προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διότι είναι πολύ σημαντικά. Αυτό το Ταμείο συνεισφέρει στους στόχους του Ταμείου Συνοχής και της πολιτικής συνοχής και επειδή χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια θα πρέπει να ισχύει αυτή η διαφάνεια και για αυτό το Ταμείο ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο κρίσης που διανύουμε. Αυτό θα βοηθούσε για να φτάσουμε σε πιο ορατά αποτελέσματα. Uh, you, um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία και καταρχήν να πω ότι στην τελευταία θητεία ασχολήθηκα με θέματα διαφάνειας σε άλλη επιτροπή και νομίζω ότι υπάρχουν τομείς όπου υπάρχουν κοινά ζητήματα προς επίλυση. Θα ήθελα να τιμήσω τον εισηγητή για μια διεξοδική εργασία και δεν, έχω, δεν αντιμετωπίζω προβλήματα με την έκθεσή του. Ο εισηγητής μίλησε για τα προβλήματα που έχουμε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με τη διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα άμα δούμε τις ε, έμπρακτες λεπτομέρειες από πλευράς agencies, κρατών μελών και ευρωπαϊκής ε, θεώρησης. Στη δική μου περιφέρεια αντιμετωπίσαμε μεγάλα προβλήματα ως προς τη διαφάνεια, δηλαδή τον τρόπο που ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις επιμεμονωμένων ε, προγραμμάτων. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε, δηλαδή να απομακρυνθούμε από την επιβολή αυτών των προαπαιτήσεων στα κράτη-μέλη και στους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό αφορά τους εμπλεκόμενους φορείς. Ένα από τα μέλη των σοσιαλιστών και δημοκρατών είπε ότι δεν πρέπει να κατονομάζουμε και να διαπομπεύουμε αλλά νομίζω ότι επιβάλλεται αυτό, γιατί εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι κυβερνήσεις, ακόμα και οι κομισιόν φταίει, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να τους εκθέσουμε. Ένας άλλος, μια άλλη συνάδελφος μίλησε για μεγάλο φόρτο. Βεβαίως είναι μεγάλος ο φόρτος γιατί έχουμε να κάνουμε με τα χρήματα των φορολογωμένων. και το κοινό πρέπει να ξέρει πώς ε, δαπανώνται αυτά τα κονδύλια. Γι' αυτό νομίζω αυτό που προτείνει ο εισήγητης, αυτά που προτείνει είναι απολύτω σωστά και κατάλληλα και συμβαδίζουν με την πρωτοβουλία διαφάνειας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα σφάλμα, εξόφθαλμο θα μπορούσα να πω γιατί μιλάμε για τη διαδικασία κατανομής πόρων όταν έχει λήξει αυτή η διαδικασία πώς αποτιμάται, τι απολογισμός γίνεται και πώς δημοσιοποιούνται τα στοιχεία. Ε, εκεί που υπολείπεται, ε, υπολείπεται στα πρώτα στάδια, διότι στην προηγούμενη θητεία ασχοληθήκαμε με το θέμα του lobbying και θα ήθελα σε αυτή την έκθεση να δω και αυτό το σκέλος, δηλαδή και στους εμπλεκόμενους φορείς και στις υπηρεσίες και στα κράτη-μέλη να έχουμε ένα κατάλογο των λόμπι που υπάρχουν για τα διάφορα project, έτσι ώστε το κοινό να ξέρει ποιος πιέζει για αυτά τα σχέδια. Θα σας εκπλήξουν ορισμένα αποτελέσματα του, η στοιχεία του καταλόγου. Ρωτώ λοιπόν τον γιατί θα μπορούσε να δεχτεί αυτή την ιδέα της δημοσιοποίησης των λόμπι και ποιοι ακριβώς ασκούν πίεση έτσι ώστε να εφαρμοστούν αυτά τα σχέδια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η έκθεση του κυρίου Τρεμόπουλου έχει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία. Έχω τη γνώμη όμως ότι δεν ανταποκρίνεται στον τίτλο της και θα πρότεινα να αλλάξουμε και τον τίτλο. Δεν νομίζω ότι τα μέτρα που προτείνονται αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το μεγάλο και υπαρκτό πρόβλημα της διαφάνειας. Γι' αυτό ίσως η έκθεση θα έπρεπε να ονομαστεί μέτρα για την ε, καλύτερη παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Από εκεί και πέρα είναι ένα πραγματικό πρόβλημα κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι πεισμένος ότι το πρόβλημα της διαφάνειας θα το αντιμετωπίσουμε με τα προβλήματα αυτά που αναφέρει ο κ. Στρεμόπουλο, που στην ουσία είναι εναρμόνιση των βάσεων δεδομένων. Από πού προκύπτει ότι αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Το λέω γιατί γενικά με ενοχλεί όταν οι συγκίσεις μας δεν έχουν και ένα τεχνοκρατικό, αν θέλετε, ένα πιο επιστημονικό υπόβαθρο. Παραδείγματο χάρη στη χώρα μου, ξέρω ότι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι οι επιτροπές, οι οποίες εγκρίνουν ή απορρίπτουν αυτά τα προγράμματα. Ποια είναι η σύνθεση αυτών των επιτροπών, ποιο τι ελέγχει, τι δυνατότητα παρέμβασης έχουν μαζικές οργανώσεις, κινήματα κτλ. σε αυτές τις διαδικασίες. Εάν αυτό δεν λυθεί, νομίζω όλα τα υπόλοιπα στην καλύτερη περίπτωση θα είναι ένας επιπλέον γραφειοκρατικός φόρτος, δεν θα λύσουν καθόλου το πρόβλημα. Δεύτερο σοβαρό πρόβλημα. Τι γίνεται όταν εντοπίζονται κρούσματα. Εγώ στην Ελλάδα δεν ξέρω μία περίπτωση, μία σας λέω, που ενώ ξέρουμε ότι γίνονται σκάνδαλα, μεγάλα σκάνδαλα, ποτέ δεν βρέθηκε κανεί στα δικαστήρια. Δεν ξέρω σε άλλε χώρε τι γίνεται. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιου είδου διαδικασίε και τέτοιου είδου πράγματα, όσο πληροφοριακά συστήματα να έχουμε, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Τελειώνοντα, θα ήθελα να πω ότι ο κύριο Τρομόπουλο είναι και λίγο γενικόλογο. Παραδείγματο χάρη, το σημείο 10 στην έκθεσή του λέει τονίζει τη σημασία τη ακριβού και έγκαιρη παροχή πληροφοριών. Ε, πόσο ακριβή και πόσο έγκαιρα πρέπει να είναι οι πληροφορίε. Ή να το πω αλλιώ, πόσο πιο ακριβή και πόσο πιο έγκαιρες από αυτές που ήδη έχουμε. Γι' αυτό λέω ότι θέλουμε συγκριτικά στοιχεία. Αλλάζουν τα project, υπάρχουν υπερβάσεις, υπάρχουν ε, ε υπερτιμολογήσεις, ε, αλλάζουν οι τιμές. Αυτά θα μπαίνουν στο σύστημα ή θα είμαστε στα αρχικά. Σημείο 12. Ε, ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν σκληρότερη στάση. Τι σημαίνει σκληρότερη, πόσο σκληρότερη, μέχρι πού να φτάσει στο σκληρότερο κτλ. κτλ. Ε, Τελειώνοντα, θα ήθελα να πω ότι όντω είναι σοβαρό το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά τα οποία ε, διακυβεύονται. Κάτι υπόθηκε να γίνουν πιο ορατά τα έργα αυτά στο, κοινό. Στη χώρα μου γίνεται αυτό. Σε όποιον δρόμο να πάτε θα έχει ταμπέλες που να λένε ότι γίνονται με χρήματα του Ευρωπαϊκού ε, Κοινωνικού Ταμείου του Ταμείου Συνοχή. Αυτό όμω δεν είναι το πρόβλημα τη διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ο κύριος Σταυρακάκης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ και εγώ τον κύριο εισηγητή, τον κύριο Τρεμόπουλο για την έκθεσή του. Είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, αδιαφυσβήτητο ότι η ενίσχυση της διαφάνειας πάνω τη στοχεύει στη χρηστή διακυβέρνηση, στη διαχείριση έργων μέσω του ελέγχου του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι να βρούμε μια και που είναι το δύσκολο σημείο, να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις προσπάθειες που κάνει η Επιτροπή μας για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση από τη μία πλευρά και τις προσπάθειες για απλοποίηση των κανόνων διαχείρισης από την άλλη. Σύμφωνα με την μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια στην πολιτική συνοχής, στις περιπτώσεις που παρατηρείται μη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσει, ε, φαίνεται να προκύπτει ότι αυτή σχετίζεται μάλλον με την έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων από πλευράς διαχειριστικών αρχών παρά την απροθυμία παροχής τέτοιων δεδομένων. Δεν θέλω να παραλάβω αυτό που υπόθηκε από τους συναδέλφους ότι ίσως δώσουμε ένα πρόσθετο ιδιαίτερο βάρος σε φορείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να το σηκώσουν. Επιπλέον, οι διοικητικέ απαιτήσει θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση αυτών των φορέων που κατά κανόνα πρόκειται για μικρού φορεί στα προγράμματα τη πολιτική συνοχή. Πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι οι απαιτήσει για την παροχή πρόσθετων στοιχείων αναφορικά με τα υλοποιούμενα έργα στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή δεν θα φτάσουν στο σημείο να αντιστρατεύονται το στόχο για απλοποίηση στη διαχείριση των διαφορετικών ταμείων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο ρόλος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να είναι καθοριστικός, αν μεριμνήσει για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους φορείς προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις όποιες πρόσθετες απαιτήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριο Πίπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή θα είναι ορόσημο για τη μελλοντική αντιμετώπιση της ε, πολιτικής συνοχής. Νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει η έκθεση αυτή πάρα πολύ λογικά θέματα και από τη δική μου πείρα έχω σας πω ότι πέρσι προσπάθησα με ορισμούς συναδέλφους να συγκρίνω τις δημοσιεύσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Ήτανε άνω κάτω. Ήταν αδύνατον να συγκριθούν τα στοιχεία αυτά. Τώρα δεν λέμε ότι θέλουμε μια ενιαία μορφή της δημοσίευσης. Όταν λέμε ότι θέλουμε τα στοιχεία αυτά να δημοσιεύονται και στα αγγλικά, τότε δεν χρειαζόμαστε αυτή την κατηγορία που λέτε, τον ονειδισμό. Είναι πάρα πολύ εύκολο τότε πια η επιστημόνες να μπορέσουν να κρίνουν τι έχει γίνει με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Ξαφνικά και εμείς ως πολιτικοί θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάποια σχέδια, να τα ελέγξουμε. Αυτή η μορφή της δημοσίευσης είναι μια μεγάλη βοήθεια και θα μπορέσει όπως και στην αγροτική πολιτική να βοηθήσει καταρχήν ε, τον έλεγχο κάποιων τομέων τη πολιτική μα, όπω το ίδιο σημαίνει και με την αγροτική πολιτική. Αυτό θα εξαρτάται από τη δική μα βούληση. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με τι ε, βασικέ ιδέε ε, τη έκθεση, μόνο με το σημείο 12 δεν συμφωνώ, δεν πρέπει να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και από την άλλη μεριά θα ήθελα να μα ενθαρρύνω να επιμείνουμε και να περάσουν τα στοιχεία αυτά στον επόμενο κανονισμό για τα διορθωτικά ταμεία. Γιατί εμεί τώρα πια είμαστε ο κοινοβούλιο μέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν εξετάσουμε τον επόμενο κανονισμό για τα διορθωτικά. Ευχαριστώ. Λίβαν Σκουτμάνης. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πράγματα. Πρώτον, Ήδη υπάρχει σήμερα ένας βαθμός ευθύνης, βαθμό ευθύνη που έχουν τα συστήματα ελέγχου, προκειμένου να λειτουργεί σωστά το σύστημα. Ξέρουμε ότι σε ορισμένες χώρες για τις εφιστάμενες δημοσιονομικές προοπτικές δεν έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή κάποια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελάχιστα κονδύλια έχουν δοθεί μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να προχωρήσουμε σε επικαλύψεις. Συμφωνώ όμω με τα όσα λέει ο συγητή για τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου. Μόνο μέσω του μέσου αυτού θα καταφέρουμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Τρίτον, α δούμε επίση το ζήτημα και από τη νομική του πλευρά. Αν καταγράψουμε τις δαπάνες πρέπει να πάνε στους ε, δικαιούχους, τους τελικούς δηλαδή δικαιούχους των ταμείων, τότε μπορεί πολύ εύκολα οι δικαιούχοι να μας πούνε ότι δεν προβλεπότανε να πρέπει να δικαιολογήσουν την ε, υφιστάμενη ε, απορρόφηση των ε, πόρων. Ότι δεν είχε προβλεφθεί αυτό δηλαδή ο σύστημα επιτήρησης από την αρχή. Αν εξετάσουμε τώρα τα agencies της υπηρεσίες, Υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία προβλέπονται για την τεχνική αρρωγή. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την οικονομική δυνατότητα για να στήσει ένα επιπρόσθετο ηλεκτρονικό σύστημα και να δημιουργήσει το δίκτυο αυτό στο οποίο αναφερθήκατε και στην ιστοσελίδα στην οποία αναφερθήκατε ώστε να μπορεί κανείς δηλαδή, να πηγαίνει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια να έχει πρόσβαση στις επιμέρους σελίδες των κρατών μελών και ε, σε όλα τα στοιχεία τα οποία θα φτάνουν σιγά σιγά μέχρι και τα στοιχεία των δικαιούχων. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα παρακολουθήσει τα ίδια ολοκληρωμένα έργα ή τα σχέδια αυτά τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη αυτή τη στιγμή που εκκρεμούν. Είναι σημαντικό επίσης και αυτό να το δούμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να ζητήσουμε από τους δικαιούχους να μας δώσουν στοιχεία για τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχή. Επίσης, γίνεται μία αναφορά σε μία μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής ε, Πολιτικής σε σχέση με μία απόφαση που έχει κάνει το ελεκτικό συνέδριο. Και φαίνεται εκεί πέρα ότι σε ορισμένες χώρες πρέπει να υπάρχουν τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα, τα οποία να καταγράφουν την ε, απορρόφηση των κονδυλίων. Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα όμως που υπάρχουν ήδη σε κάποια κράτη-μέλη δεν λειτουργούν σωστά και σε ορισμένε περιπτώσεις έχουν μπλοκάρει την απορρόφηση των κονδυλίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όντως δημιουργείται επιπρόσθετος φόρτος αν τα συστήματα αυτά εφαρμοστούν και δεν λειτουργήσουν στην πράξη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σίγουρα το διαδίκτυο, θα πρέπει να εξετάσουμε και τα ολοκληρωμένα project, τα ολοκληρωμένα προγράμματα και βάσει αυτό να καταφέρουμε να πάρουμε πληροφορίες με πιο εύκολο τρόπο από τα agencies και έπειτα να αποφύγουμε να θέσουμε όλο το φόρτο στους δικαιούχους, γιατί θα έχουμε πολλά νομικά προβλήματα και επίσης να έχουμε και μία προσωρινή μεταβατική περίοδο, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε μία νυχτή από τη μία μέρα στην άλλη να επιβάλλουμε τόσο αυστηρές διαδικασίες ε, διαφάνειας. Ευχαριστούμε πολύ. Eh, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Καταρχάς, να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ καλή του αυτή έκθεση. Και θεωρώ ότι ε, οι παρεμβάσεις των ε, συναδέλφων θα εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο την συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι κατά την άποψή μου εδώ πέρα αναφερόμαστε σε ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι έχουμε πει μέχρι στιγμής. Το ζήτημα αυτό της πληροφόρησης των πολιτών πρέπει να προωθηθεί στην πράξη και να μην ε, επαφιόμαστε απλώς σε ωραίες φράσεις όπως ε, η διαφάνεια. Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι πολίτες να αισθάνονται ότι ε, εμπλέκονται περισσότερο σε αποφάσεις που λαμβάνονται, να λαμβάνουν την απαραίτητη ενημέρωση και να μην αισθάνονται ότι όλες οι αποφάσεις και ότι όλη η ενημέρωση τελικά έρχεται από ένα απόμακρο θεσμικό όργανο. Άλλωστε, οι επικρίσει που ακούμε πάρα πολύ συχνά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι είναι πάρα πολύ μακριά από τον Ευρωπαίο πολίτη. Θεωρώ λοιπόν ότι μα δίνεται εδώ πέρα μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στου Ευρωπαίους πολίτες. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσει. Πρώτον, πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε να μην δίνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε πάρα πολλέ μελέτε διαβάζουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε βομβαρδίζονται από πάρα πολλέ διαφορετικέ πληροφορίε σε καθημερινή βάση. Οι πληροφορίε αυτέ μπορεί να είναι οι ειδήσει, ένα άρθρο το οποίο διαβάζουν στην εφημερίδα κτλ. και μετά από δύο ημέρες από τη στιγμή που θα λάβει κανείς μια πληροφορία θα καταφέρει να διατηρήσει ελάχιστες από τις πληροφορίες αυτές που του ε, έχουν δοθεί. Έχει υπολογιστεί ότι σε ένα σύνολο χιλίων πληροφοριών ο πολίτης μπορεί μετά από δύο μέρες να διατηρήσει 40 μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές ε, δίνει πολύπλοκες και δυσνόητες πληροφορίες προς τον ε, Ευρωπαίο πολίτη, με αποτέλεσμα ο πολίτης τελικά να μην καταγράφει καθόλου τις πληροφορίες αυτές, να τις απορρίπτει. Μπορεί κανεί να μιλάει για διαφάνεια στην περίπτωση αυτή, αλλά οι πληροφορίε οι οποίε δίνονται τελικά στου πολίτε δεν είναι ενδιαφέρουσε για τον πολίτη. Δεν μπορεί ο πολίτη να τι επεξεργαστεί τι πληροφορίε αυτέ. Και γι' αυτό το λόγο συμφωνώ με τον οσηγητή ότι θα πρέπει οι πληροφορίε που δίνουμε να είναι σαφεί και απόλυτα συγκρίσιμε από τη μία χώρα στην άλλη. Ουσιώδει δηλαδή πληροφορίε, ξεκάθαρε, Μία ακόμα παρατήρηση θέλω να κάνω. Θεωρώ ότι η έκθεση είναι απόλυτα ικανοποιητική όσον αφορά τα μεγάλα προγράμματα, τα μεγάλα σχέδια. Τις σημαντικές δηλαδή επενδύσεις, όπου οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται σε επίπεδο κράτους μέλους, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και στην περίπτωση όμως αυτή δεν έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Βάσει ποιο στοιχείων, βάσει ποιο δεδομένων οι Βρυξέλλες αποφασίζουν για τα μεγάλα αυτά προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για παράδειγμα, δίνει πάρα πολλά στοιχεία και πληροφορίες προτού καν να αποφασίσει ποια δάνεια θα πρέπει να δοθούν σε συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα. Ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτό το παράδειγμα. Υπάρχει τουλάχιστον ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που δίνει περισσότερες πληροφορίες και μάλιστα εκ των προτέρων. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω το συνάδελφο και να υποστηρίξω ότι συνεχίζει μία ιδιαίτερα καρποφόρα συζήτηση που άρχισε πέρσι με μία εξίσου σημαντική έκθεση του συναδέλφου ε, Jean-Marie ο οποίος μιλούσε για multi-level governance. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η πολύπλευρη διακυβέρνηση αν δεν υπάρχει διαφάνεια και διάλογος. Η διαφάνεια είναι ε, πρόκριμα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την χρηματοδότηση αυτή. Δεν μπορεί να υπάρχει προβλεψιμότητα σε περιφερειακό επίπεδο αν δέξουμε για τι περιφερειακή διάσταση μιλάμε. Νομίζω ότι η διαφάνεια είναι ύψης της σημασίας ως προς την ε, αλλαγή της πολιτικής μας, κάτι το οποίο αφορά την ΚΑΠ και την περιφερειακή πολιτική. Και τώρα επανέρχομαι στη δική μου χώρα θα ήθελα να πω δυστυχώς ότι υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη διαφάνειας ως προς την περιφερειακή μας πολιτική, ώστε μας υποδείξατε πέρσι να προβούμε σε μια περιφερειακή πολιτική έτσι ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα κονδύλια μας. Επειδή λοιπόν υπήρχε πλήρης έλλειψη διαφάνειας, αλλάξαμε την περιφερειακή μας ε, οικοδόμηση, χωρίς όμως να μιλήσουμε με πολιτικά κόμματα και κοινωνικούς φορείς. Και η γερουσία μας ε, προέβαλε ένα νόμο για το, την περιφερειακή μεταρρύθμιση, χωρίς να υπάρχει καμία διαφάνεια και προγενέστερος ε, διάλογος. Γιατί μιλάμε για διαφάνεια τη στιγμή που στη ε, Ρουμανία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία διαφάνεια στο δημόσιο φορέ. Και οι υπάλληλοι δεν μπορούν να κοινοποιούν στοιχεία τα οποία επιτρέπονται ρητός. Και δυστυχώς ο, οι, πολλές φορές υπεύθυνοι υπουργείων λένε ότι δεν έχουμε άδεια να κοινοποιούμε πληροφορίες. Δεν το λέω αυτό γιατί πρόκειται για τη χώρα μου, αλλά επειδή πιστεύω ότι δεν πρέπει να προβάλλεται σαν μια πάγια πολιτική. Θα ήθελα να τιμήσω το συνάδελφο και νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε ε, κριτήρια και επίσης ε, συνοχή για τα 27 κράτη καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα υποχρεωτικά και με κυρωτικές ε, ρήτρε τη στιγμή που παραβαίνονται τα κριτήρια. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα αφήσουμε τόπο στις καταχρήσεις και στις απάτες. Ο Ευρωπαίος πολίτης δεν θα μπορεί να ξέρει από πού προέρχονται τα πολιτικά ευεργετήματα της συνοχής για το σχολείο του, για το νοσοκομείο του, για όλες τις δημόσιες υποδομές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια έτσι ώστε να έχουμε και την υποστήριξη του μέσου Ευρωπαίου πολίτη. Ευχαριστώ. Ε, very Προτού δώσω το λόγο στον τελευταίο μιλητή, Πρέπει να σας πω ότι κανένας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα συμβούλευε ποτέ ένα κράτος μέλος πώς να προχωρήσει με την εθνική πολιτική όσον αφορά τα διαφορετικά ταμεία. Πρόκειται για μια καθαρά εθνική πολιτική. Ε, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω η διαδικασία της, οι διαδικασίες της διαφάνειας είναι πάρα πολύ καλές και βοηθούν στη διακυβέρνηση, στη χρηστή διακυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής διανύουμε μία περίοδο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου θα πρέπει, με βάση την οποία θα πρέπει να πλουστέψουμε τις διαδικασίες πρόσβασης στα ευρωπαϊκά ταμεία. Θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 9 της ε, πρότασης ψηφίσματος, όπου τονίζεται η πιθανότητα να απλουστεύσουμε το πλαίσιο αυτό και έτσι ώστε οι ευεργετούμενοι να έχουν καλύτερη πρόσβαση και για να μειωθεί και ο διοικητικός φόρτος. Θα ήθελα και αυτή η έκθεση να εγγραφεί σε αυτά τα πλαίσια, δηλαδή να απλουστεύσουμε την διαδικασία πρόσβασης και να μην έχουμε έναν επιπρόσθετο διοικητικό φόρτο. Δηλαδή να μην υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία για ε, ορισμένα κράτη. Ελπίζω λοιπόν να γίνει αυτή η απλούστευση ως προς τη ε, διοικητική διαδικασία και το διοικητικό φόρτο, διότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μου γίνεται μία διαβούλευση. Εμείς δεν έχουμε τις περιφέρειες που δρούν σαν διοικητική μονάδα και γι' αυτό θα πρέπει να διανύσουμε ε, αυτή τη διαδικασία και το δύσκολο δρόμο για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ε, διοικητικής υποδιέρεσης της χώρας μας και σε επίπεδο περιφερειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Φίσερ, σύντομα ενδεχομένω θα μπορούσε να απαντήσετε στα σημαντικότερα ερωτήματα που ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πίτερ Φίσερ από το Τμήμα Ενημέρωσης της ε, DG Regio. Σας ευχαριστούμε για την ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση. Όντως καταγράφεται και τις προσπάθειες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους δικαιούχους σε όλα τα κράτη-μέλη. Πολλές ε, από τις ε, συστάσεις οι οποίες προτείνεται κατευθύνονται στον δρόμο που έχει υποδείξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αναφέρεστε βέβαια και στο δίκτυο Inform Ορισμένες από τις συστάσεις μπορούν να εφαρμοστούν πιο εύκολα από άλλες. Πρόθεση της δεύτερης γλώσσας, τον υπάρχουν ε, περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι ευρωβουλευτές που είπαν ε, ότι υπάρχει ήδη ένας κανονισμός αυτή τη στιγμή ενισχύει, βάσει του οποίου ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι περαιτέρω. Αυτό που προσπαθούμε όμως να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη ασκώντας πίεση και προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές μέσω του υφιστάμενου δικτύου. Έχουμε κάποιες πολύ καλές ιστοσελίδες τις οποίες ε, έχουμε χρησιμοποιήσει στις συνεδριάσεις που έχουμε κάνει σε διάφορες χώρες, όπως την Λιθουανία, την Ουγγαρία, σε κάποιες περιφέρειες της Αυστρίας επίσης. Βλέπετε εκεί πέρα ιδιαίτερα πολύπλοκα προηγμένα συστήματα. Ορισμένες φορές έχουμε μάλιστα και τους καταλόγους των δικαιούχων που έχουν ανταποκριθεί στις ελάχιστες απαιτήσει, αλλά έχουμε και άλλα στοιχεία στα πλαίσια των ιστοσελίδων αυτών οι οποίες θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα προσβάσιμες και αναφέρομαι στο στοιχείο αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αυτά γιατί καθιστούν το σύνολο της περιφερειακής πολιτικής πολύ πιο ορατό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωνόμαστε μόνο σε κάποια εργαλεία, σε κάποια όργανα, αλλά να δούμε το σύνολο των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα επίσης να φερθώ σε μία παρατήρηση που ακούστηκε πριν από λίγο. Ορισμένες συστάσεις πρέπει να μπουν στον κανονισμό που θα αφορά την περίοδο 2014-2020, ενώ υπάρχουν ε, κάποιες άλλες συστάσεις που ουσιαστικά ζητούν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον κατάλογο των δικαιούχων και όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των ιστοσελίδων. Θα είμαι σε επαφή μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες πάντως. Ε, Μιχάλη, θα θέλατε να ξαναπάρετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για, τις, ε, και για τα καλά λόγια και για τις ε, παρατηρήσεις που προφανώς είναι χρήσιμες. Είδα ότι υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Εκείνο όμως που θα ήθελα να ε, τονίσω είναι ότι οι χώρες δεν έχουν ε, τον ίδιο βαθμό καταγραφής αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων και των δυνατοτήτων και των πληροφοριών. Προφανώς σε κάποιες χώρες αρκετά από αυτά που λέμε να εφαρμόζονται. Οι σεφορείς, υποδείξαμε κιόλα ποιοι. Αλλά έχει σημασία να γίνει κάτι ενιαίο. Είδατε την αγωνία ε, συναδέλφων που εκπροσωπούν χώρες της περιφέρειας, όπου εκεί δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι γνωρίζουν οι πολίτε, οι ενδιαφερόμενοι, ε, ποια προγράμματα υπάρχουν ποιε προθεσμίε τρέχουν, δεν έχουν δηλαδή εκείνη την πληροφόρηση και τη βοήθεια ώστε έγκαιρα να κινηθούν. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο να κοιτάμε τι ταμπέλε όταν έχει γίνει ένα έργο, αλλά εδώ τονίζουμε και την ανάγκη να μαθαίνουν οι ενδιαφερόμενοι ακόμη και πριν την απόφαση για τη χρηματοδότηση κάποιων έργων. Άρα αυτή η μεταβλητότητα στις συνθήκες σε κάθε χώρα δεν επιτρέπουν όπως υπόθηκε την πλήρη σύγκριση του τι συμβαίνει σε κάποια χώρα. Το ακούσαμε από, από συνάδελφο ότι τα πάντα είναι άνω, άνω κάτω στις διάφορες χώρες. Λέμε κομψά για διαφορετικές διοικητικές ικανότητες και πολιτισ, πολιτιστικές παραδόσεις. Να σας πω και η εμπειρία έρχεται και από τη δικιά μου χώρα ότι αυτές οι δυσκολίες είναι υπαρκτέ. Και ε, όπου από ό,τι μας δόθηκε ευκαιρία να δούμε και σε άλλες χώρες υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες. Δεν μιλάμε για παραπάνω γραφειοκρατία, κανείς δεν τη θέλει. Αλλά για διευκόλυνση αυτών των στοιχείων που ήδη υπάρχουν. Δεν μπορεί η Επιτροπή να περιορίζει το ρόλο της στο να λέει κάποια ενδεικτικά πρότυπα και κατευθύνσεις. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες πιο λεπτομερείς πληροφορίες, να προσδιορίζονται δηλαδή η δομή, η μορφή, το περιεχόμενο των πληροφοριών που κάθε κράτος πρέπει να παρέχει. Αυτό το ενιαίο προσπαθούμε, ούτω ώστε να υπάρχει και ισότητα στην πληροφόρηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών και γι' αυτό και πρέπει να είναι, υπάρχει αυτή η διαφάνεια και στο πριν και στο μετά. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές και με αυτή την έννοια θα το δούμε και στη συνέχεια τις παρατηρήσεις που έγιναν θα προσπαθήσουμε να τις πάρουμε υπόψη. Βέβαια όταν είναι συγκρουόμενες ε, θα αποφασίσει το σώμα. Για παράδειγμα στο άρθρο 12 που σχολιάστηκε για την κατονομασία και ονειδισμό ε, προφανώς υπάρχει ένα θέμα. Πάντως η δικιά μου εμπειρία λέει ότι ε, οι, οι, οι συνθήκες και η συζήτηση που γίνεται γύρω από την Ελλάδα και τα στοιχεία τα οποία παρουσίαζε πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση έγκαιρα και όχι όταν διονγκωθεί το πρόβλημα. Θέλουμε δηλαδή να προλάβουμε και όχι να έρθουμε μετά να κάνουμε κριτική. Γι' αυτό και υποστηρίζω αυτή την, αυτό το, το άρθρο, αλλά το σώμα θα αποφασίσει για το αν θα πρέπει να προχωρήσει παραπέρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 24 Μαρτίου στις 6 το βράδυ είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Όσοι επιθυμείτε λοιπόν να υποβάλλετε τροπολογίες παρακαλώ πολύ μέσα στην προθεσμία αυτή να το κάνετε. Και πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποίησαμε τρεις φορές παραπάνω χρόνο από ό,τι προβλεπόταν στη μερίσια διάταξη για το ζήτημα αυτό και συμφωνώ μαζί σας ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε ελάχιστο πλέον χρόνο για το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Σας ζητώ λοιπόν να δείξετε απόλυτη πειθαρχία με τον χρόνο. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το ζήτημα το οποίο θα μας παρουσιάσει συντομότατα ο Πέτρου Λούχαν. Θα ήθελα να σας πω ότι μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα διότι είναι ένας από τους όρους εκ των ουκ άνευ για να φτάσουμε σε αυτή τη συνοχή σε όλα τα επίπεδα. Πρόκειται για μία ερώτηση που αφορά το πρόσωπο της πολιτικής ε, συνοχής που κινείται σε τρία σκέλη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συγκρίνουμε αυτή τη διαδικασία με την βαθμιαία, ένα και μεγαλύτερη μάλλον σημασία του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε αυτές τις τρεις διαστάσεις την οικονομική με την κοινωνική καθώς και την εδαφική, όπως ορίζει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Και θα πρέπει να αναλάβουμε, να λάβουμε τις ε, κατάλληλες αποφάσεις έτσι ώστε να ακουστεί και η φωνή του Ευρωπαίου πολίτη. Δηλαδή πέρα από την οικονομική και κοινωνική πολιτική ε, συνοχής να ασχοληθούμε και με την εδαφική συνοχή. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε μία ιεράρχηση προτεραιοτήτων από πλευράς περιφερειακής θεώρησης, διότι αυτό προσλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία για να ε, λάβουμε κοινοτικές αποφάσεις. Το Ευρωβαρόμετρο το Φεβρουάριο του 2010 σε σχέση με την ε, κοινή γνώμη μας δείχνει ότι υπάρχουν δύο βασικές ανησυχίες. Δηλαδή, ο πληθωρισμός και η οικονομική κατάσταση. Τι σημαίνει για να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να επιλύσουμε πρωτίστως τα προβλήματα του πολίτη. Έχουμε το θέμα της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας, τη συζήτηση της στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, να ορίσουμε τις τομεακές πολιτικές και να δούμε πώς θα φτάσουμε στην αύξηση της ε, οικονομικής ε, ανταγωνιστικότητας επιλύοντας τα οικονομικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας προτείνω ορισμένες ε, πρωταρχικές σκέψεις, ένα προήμιο σκέψεων, και μετά από πολλές διαβουλεύσεις αποφάσισα να σας μιλήσω για τις προοπτικές ε, της ε, ανάπτυξης του οικονομικού, της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε και τις επενδύσεις στις υποδομές, στις μεταφορές, στην εκπαίδευση και ούτω καθεξής θα πρέπει να προσδώσουμε σημασία στα 12 κράτη τα οποία προσχώρησαν αργότερα και να δούμε ποια θέματα, ποιες πτυχές ε, είναι ύψης της σημασίας έτσι ώστε να προγραμματίσουμε την περίοδο 2014-2020. Στην αρχή έχω ορισμένες πηγές πληροφοριών και έργα. Αναφέρομαι σε ψηφίσματα και εκθέσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης που έχουν συνταχθεί, ιδιαίτερα σε σχέση με την εδαφική συνοχή. Μετά βλέπετε τον τρόπο εκτίμησης αυτών των μέτρων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων και για να δούμε πώς εφαρμόζεται η πολιτική σύνοχης, έτσι ώστε να προβούμε και σε μια βελτίωση και απλούστευση διαδικασιών, να έχουμε καλύτερο συντονισμό, καθώς και ευελιξία των ταμείων. Επίσης έχουμε την έκθεση του 2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία άνοιξε μία σειρά από ερωτήματα και οι επόμενες δύο εκθέσεις έχουν αποσαφηνίσει την κατάσταση που ισχύει στον τομέα της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια των καινοτομιών και της έρευνας. Η έκθεση Μπάρκα είναι καθοριστικής σημασίας για την αναθεώρηση της ε, περιφερειακής ε, πολιτικής. Έχει σημασία να δούμε πώς ε, μπορούμε να ανταποκριθούμε και στον παγκόσμιο οικονομικό ιστό. Πέρα από τα στοιχεία και τις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε και πληροφορίες από την ΕΤΕ έτσι ώστε να έχουμε μία σαφή εικόνα για τις επιπτώσεις της πολιτικής συνοχής στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε ποια, ε, μάλλον πού ε, αποτάθηκαν και πού ποια στοχοθέτηση είχαν ε, τα κονδύλια και τα ταμεία και στην περίπτωση των επενδύσεων από πλευράς ΕΤΕ βλέπουμε ότι ότι τα 12 κράτη που προσχώρησαν αργότερα έχουν προβεί σε σχέδια ε, δάνειοδοτήσεων μέση της ΕΤΕ. Βλέπετε ποιες είναι οι άμεσες ανάγκες σε περιφερειακό επίπεδο και βλέπουμε ότι η οικονομική ε, συνοχή μπορεί να επιτευχθεί ίσως καλύτερα και πιο γρήγορα από ό,τι νομίζαμε. Επίσης, μας ενδιαφέρουν οι θέσεις των παγκοσμίων φόρουμ και αυτό που έχει σημασία είναι πώς ορίζουμε την παραγωγικότητα σε κάθε κράτος μέλος. Δηλαδή, έχουμε 16 πυλώνες εδώ. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ε, μπορούμε να συνεισφέρουμε στην αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η έκθεση για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πλαίσιο της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοίξει τις πόρτες της και να κοιτάξει προς τα έξω. Ως προς τη μεθοδολογία, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σχέση μεταξύ πολιτικής πολιτικής, της πολιτικής πολιτικής του περιεχομένου και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σημασία να δούμε και την ανάγκη ενίσχυσης και διατήρησης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας μέσω της κατάλληλης υποδομής που έχει τα κατάλληλα, τα ανάλογα χαρακτηριστικά σε όλες τις περιφέρειες η αφετηρία θα είναι η ανάλυση των προτεραιοτήτων που έχουν προσδιοριστεί από τα 12 κράτη-μέλη μέσα στα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς. Σημασία έχουν και τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς και τα projects ε, με βάση τα οποία η ΕΤΕ προέβησε δανειοδοτήσεις. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι περιφέρειες της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης έχουν πληγεί περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να δούμε πώς θα οικοδομήσουμε το μέλλον μας έτσι ώστε να έχουμε κοινές πολιτικές σύνοχης με τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την προώθηση βασικών προτεραιοτήτων για κάθε περιφέρεια. Γιατί υπάρχει άνηση, υπάρχουν άνηση, υπάρχει άνηση ανάπτυξη και διαφορετικές ανάγκες. Επίσης θα πρέπει να γίνει η σωστή κατανομή των Ταμείων Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ανάλογα με τις ανάγκες των περιφερειών. Επίσης, θα δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ε, προώθηση της οικονομικής συνοχής και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλους και στον τομέα της ε, υποδομής, των ε, κοινωνικών προδιαγραφών και της εκπαίδευσης. Αυτό που έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το έγγραφο εργασίας για να συνταχθεί στη συνέχεια αυτή η έκθεση που είναι πολύ σημαντική για την ε, πολιτική συνοχής, μια βιώσιμη πολιτική συνοχής και γι' αυτό χρειάζεται ανταλογή απόψεων όπου όλοι θα είναι κοινωνοί και αναμένω τα σχόλιά σας. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ και πάλι να είστε πολύ σύντομοι. Θα έχουμε και στο μέλλον την δυνατότητα να συζητήσουμε την έκθεση αυτή. Λάμπερ Βανίστερόι. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να υποβάλω κάποιες ιδέες. Ίσως θα πρέπει κάπως να οριοθετήσουμε λίγο τη συζήτηση αυτή τη στιγμή και να αναφερθούμε στα βασικά ερωτήματα που όντως βασικό ερώτημα είναι η επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και δαφικής συνοχής στα πλαίσια ενός ε, νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να επιλέξουμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και θα μπορέσουμε να αναλύσουμε περισσότερο το ευρωπαϊκό μοντέλο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο Αλληλεγγύη στο ευρωπαϊκό μοντέλο συνοχής, το οποίο έχει συμβάλει πάρα πολύ στην ανάπτυξή μας τα τελευταία 20-25 χρόνια. Και βάσει του μοντέλου αυτού θα πρέπει να ταινίσουμε το μέλλον και να δούμε πώς θα μπορούσε το μοντέλο αυτό να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτή η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά για τη δημιουργία της Ευρώπης που εμείς θέλουμε. Μια Ευρώπη ισορροπημένη, με συμμετρία. Στο γενικό λοιπόν αυτό επίπεδο πιστεύω θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε σημαντικά και συμφωνώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τις μελέτες του ΩΣΑ οι οποίες έχουν ασχοληθεί με πολύ συγκεκριμένε πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης. Αναφέρονται επίσης και στις μακροπεριφέρειες οι μελέτες αυτές και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαν οι μελέτες αυτές να έχουν αντίκτυπο στην εξέλιξη των περιοχών αυτών τα επόμενα χρόνια. Και μία τελευταία παρατήρηση. Μιλήσαμε για υποδομές. Οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές, σαφώς. Αλλά ας δούμε τα TENS, τα διευρωπαϊκά δίκτυα δηλαδή όσον αφορά τις υποδομές, αλλά και όσον αφορά τη, τα ευρυζωνικά δίκτυα. Βλέπουμε ποιες είναι οι αλλαγές που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε και να προσαρμοστούμε στα πλαίσια των ΤΕΝ. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα καταφέρουμε να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας για μια περίοδο μετά το 2030 και ας δούμε πώς θα καταφέρουμε ουσιαστικά να περάσουμε όλες τις ιδέες αυτές στην τελική έκθεση την οποία εσείς θα υποβάλλετε. Ευχαριστώ. Hm. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λούχαν για τι ε, προκαταρικέ σα σκέψει για την έκθεση και την ε, πολιτική Συνοχή που όπω είπε και ο κ. Φανής Λεωρή θα μα αποσχολήσει πολύ στο μέλλον. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο κ. Λούχαν ότι όσον αφορά την αξιολόγηση πολιτική ε, συνοχή, θέλει να συγκεντρώσει την προσοχή του στι 12 τελευταίε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει επίση ότι το θέλει αυτό γιατί η πολιτική συνοχή εκεί ε, οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες όσον αφορά τις υποδομές. Με αυτό νομίζω θα είμαστε όλοι σύμφωνοι και μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι η πολιτική συνοχή είναι μια από τις πιο επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης μέχρι στιγμής. Αυτό καλό, αλλά εκεί που δεν συμφωνώ είναι ότι οι περιφέρειες αυτών το 12 χωρών επλήγησαν περισσότερο από οποιοδήποτε από την κρίση και είναι πιο πολύ εκτεθειμένε στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικότερα. Ας πάρουμε τη Γερμανία. Εγώ είμαι από το Βερολίνο. Το Βερολίνο, όσον αφορά τη σειρά των 16 ομοσπονδιακών κρατηδίων, στην οικονομική ανάπτυξη βρίσκεται τελευταίο. Όσον αφορά τις επιπτώσεις οικονομικής και χρηματοπιστικής κρίσης, λένε όλοι ξεκάθαρα ότι εμείς επλήγημεν λιγότερο σαν πόλη του Βερολίνου. Γιατί τις μεγαλύτερες απώλειες ε, υπέσαν οι περιφέρειες οι οποίες έχουν πάρα πολύ βιομηχανία και οπωσδήποτε το Βερολίνο δεν ανήκει σε αυτές. Αυτές οι περιοχές είναι που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μεταφορές επιχειρήσεων, κλεισίματα επιχειρήσεων, αύξηση της ε, ανεργίας και η αποδοτικότητα της ε, βιομηχανίας μειώθηκε. Ότι η επιπτώση λοιπόν της οικονομικής κρίσης στη Γερμανία δεν ήταν τόσο υψηλές οφείλεται στο γεγονό ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βοήθησε με εκατοντάδες δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επιπτώσεις από τα προγράμματα αυτά θα μας απασχολήσουν όμως προσεχώς. Θα τις μπροστά μας τις επιπτώσεις. Δεν πρέπει λοιπόν να λέμε ότι εκείνοι που ήταν ισχυροί ήταν ισχυροί και οι άλλοι παραμένουν αδύναμοι και ότι η πολιτική συνοχή έχει σαν στόχο μόνο να προωθήσει εκείνους που είναι αδύναμοι. Ακριβώς λόγω της επίκαιρης κατάστασης σήμερα νομίζω ότι η εικόνα που δίνεται δεν είναι σωστή και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε η πολιτική συνοχή σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στρέφομαι προς τον κύριο Όλμπριχ και λέω ότι η μόνη ε, χώρα η οποία ε, παρουσίασε οικονομική ανάπτυξη το τελευταίο χρόνο ήταν η Πολωνία, που και αυτή βρίσκεται όμως στα περιθώρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεωγραφικά. Πάντως εντάξει, το θέμα θα το συζητήσουμε διαμακρόν αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ζωπολ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προβασκευτική εργασία που επιτέλεσε και μας δίνει κάποιες βάσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά την άγουσα που θέλει να ακολουθήσει, έχω δύο προβλήματα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω στο σύντομα. Η πρώτη μου παρατήρηση αφορά αυτή του προλύσαντα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να βασιστούμε με τα μέτρα μας στη μελέτη των 12 τελευταίων χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η πολιτική συνοχή αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στις 12 τελευταία ενταχθήσεις χώρες. Μια δεύτερη παρουσίαση, επίσης πολύ σύντομα. Θεωρώ ότι το θέμα της ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Άνωσης δεν τοποθετείται σωστά, παραμένει ασαφές και γενικό. Σαν να πρόκειτο για θέμα της ανταγωνιστικότητας, προσχάνει της ανταγωνιστικότητας, ενώ πρόκειται για ένα στόχο σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο μου φαίνεται ότι θα πρέπει να προσανατολιστεί προς την αηφόρο ανάπτυξη. Υπάρχει ένα συσχετισμό μεταξύ της αναβοσικότητας και της αηφόρου ανάπτυξης. Και μέσα στα πλαίσια του αηφόρου ανάπτυξης ίσως δεν εξετάσουμε σωστά το θέμα της αναβοσικότητας. Παραδείγματο χάρη, δεν μπορούμε να φανταστούμε αύξηση των υποδομών στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια χωρίς να εξετάσουμε το θέμα των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου ή την διατήρηση της βιοπικιλομορφίας. Θα πρέπει λοιπόν να τοποθετηθούμε στο σωστό πλαίσιο και το θέμα της αγωνιστικότητας θα πρέπει να εξεταστεί και αυτό μέσα στα πλαίσια που σας προανέφερα. Ευχαριστώ. Ραμόνα Μανέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Λουχάν για την έκθεση αυτή, διότι πολιτική συνοχής και ανταγωνιστικότητας είναι δύο από τους πυλώνες που ορίζουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Χρειάζεται συντονισμός σε επίπεδο όλων των κρατών μελών μέσα στα πλαίσια της συμμετοχής, της συμπερίληψης και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η αύξηση της παραγωγικότητας η καλύτερη εκπαίδευση και ένα εργατικό δυναμικό το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις προκλήσεις της ε, σύγχρονης τεχνολογίας. Γι' αυτό υπάρχει και αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των δύο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα χωρίς την απαραίτητη πολιτική συνοχή. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει στην έκθεση να υπογραμμιστεί ο σύνδεσμος, ο δεσμός μεταξύ αυτών των δύο αξώνων δηλαδή να ισχύσει μια γενική πολιτική συνοχής μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Μιλάμε για επενδύσεις στον τομέα των υποδομών, έτσι ώστε τα 12 κράτη-μέλη που προσχώρησαν αργότερα να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μια πολιτική συμπερίληψης όπου να λαμβάνουμε υπόψη και τον ε, κοινωνικό και τον οικονομικό ε, άξονα, ιδιαίτερα για τις περιφέρειες που έχουν ε, μεγαλύτερη ανάγκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λουχάν για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία, διότι συζητάμε για άλλη μία φορά μεγάλα θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η πολιτική συνοχής, καθώς και το μέλλον αυτής. Και θα ήθελα να πω στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και των κλιματικών αλλαγών, και με βάση τις δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη, και με βάση βεβαίως τη μεγάλη οικονομική κρίση υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές και ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε να μειωθούν αυτές οι ανισότητες γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένα πρότυπο το οποίο να είναι ε, άξιο να το ακολουθήσει κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να συζητήσουμε για τις υποδομές, διότι το λέμε για άλλη μία ακόμα φορά, είναι ένα θέμα το οποίο μας, ε, ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα και θα πρέπει να καταβληθούν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάποια σχόλια να κάνω και να εκφράσω και κάποιες ανησυχίες. Πολλές φορές ε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα με κάποια κείμενα Παραδείγματο χάρη έχουμε μια έκθεση με τίτλο που λέει «Πραγματοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφιακής συνοχής» εκ των άνευ της διεθνούς Αυτό όμως το θέμα που τίθεται είναι πραγματικά ένας όρος. Και τι όρος. Για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Όχι. Είναι ένας όρος ε, για μια ανταγωνιστική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ναι, αλλά όχι όμως για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Γιατί η συνοχή δεν είναι ένας όρος για την διεθνή ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να μην εκφράζουμε τα πράγματα περιτά και εσφαλμένα. Δεύτερη παρατήρηση. Θα ήθελα να προτείνω στον συνάδελφο Λουχάν να μην γράφει ε, εκθέσεις που κανένας ποτέ δεν πρόκειται να διαβάσει. Σας το λέω εκ των προτέρων, ότι εμείς είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν ένα ντοκτορά για την πολιτική συνοχής. Αυτό που θέλουμε είναι μια πολιτική θέση, ξεκάθαρη για το θέμα. Αν αρχίσουμε να αναλύουμε τι θα γίνει και ποιες είναι οι σχέσεις που υπάρχουν εδώ μεταξύ τους, θα υπάρχουν αυτονόητα πράγματα. Στη συνθήκη λέγεται ξεκάθαρα ότι το θέμα της συνοχής είναι απολύτως απαραίτητο για να υπάρχει καλός ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, εάν εμείς προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε, σημαίνει ότι δεν χρησιμεύεται τίποτα η συνθήκη που το προϋποθέτει. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν κατά πόσον αυτές οι τρεις στοιχές της συνοχής έχουν ε, αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το θέμα που τίθεται. Πρόκειται δηλαδή μόνο για την εξισορρόψη των εσωτερικών ανισορροπιών. Ας μην ξεχνάμε ότι η πολιτική τη συνοχή καλύπτεται από δύο πτυχές, δηλαδή σύγκληση και ανταγωνιστικότητα των περιφερειών. Είναι αυτονόητα τα πράγματα λοιπόν. Άμα λέμε ότι η συνοχή είναι και η σύγκληση και η ανταγωνιστικότητα, από εκεί και πέρα έχουμε ξεκάθαρο πολιτικό θέμα για την Κομισιόν κατά πόσο η πραγματικότητα αυτών των διαφορετικών πτυχών είναι απαραίτητη για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι ή όχι. Εάν ναι, τη χρειαζόμαστε. Αλλιώς είναι περιττό. Και χρησιμεύει μόνο ε, στην εξίσωση των εσωτερικών διαφορών. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται, αλλά αυτό είναι το θέμα. Δεν χρειάζεται να γράψουμε 120 σελίδες, μπορούμε να πούμε ναι, αλλά για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να κάνουμε το ΑΒΓ και να πούμε ακριβώ τι πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια τη πολιτική συνοχή για να μπορέσει η πολιτική αυτή να η καταστεί σημαντική για την αγωνιστική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμαστε στην οικονομική, στην κοινωνική και στην εδαφική πλευρά. Αναφερόμαστε την περίοδο μετά από το 2014 και θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε για το τομέα αυτό, ούτως ώστε η πολιτική συνοχή να είναι πραγματικά απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον που εδώ αναφέρομαστε στο βαθμό ανταγωνιστικότητας. Πώς αναλύεται όμως η ανταγωνιστικότητα, βάσει ποιων κριτηρίων, τι πρέπει να γίνει για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ε, κατακλείδη. Θα πούμε αυτό που είπε ο Λομπέρ. Δηλαδή, να περιοριστήσουμε σε ένα πολιτικό μήνυμα Πρόκειται για προφανή θέματα εδώ. Θα πρέπει να πούμε τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια, τι πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε η οικονομική, η κοινωνική και εδαφική συνοχή μπορεί να έχει επίδραση στην ανοιχτικότητα της Ένωσης. Και τέλος. Ε, προειδοποιώ δεν πρέπει να αναφέρουμε στα 12 νέα κράτη-μέλη, γιατί αν μιλάμε για τα 12 νέα κράτη-μέλη δεν θα υπάρχει πια συνοχή. Συνοχή αφορά όλη την Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε για την συνοχή όλη της Ένωσης, όχι τη συνοχή των 12 νέων κρατών μελών. Υπάρχουν βέβαια κάποιες καλές ιδέες από την έκθεση, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που είναι διαθέσιμες, αλλά τώρα να προσπαθήσει κανένας να αναθεωρήσει σε 10 σελίδες πριν τα βιβλία είναι υπερβολικό. Συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους και χαίρομαι για αυτή την ε, πρωτοβουλία, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στο εδαφικό, στην πολιτική συνοχή, όπως είπε και ο κύριος Όλμπριχτ. Ξέρουμε ότι οι περιφερειακές ανισότητες έχουν επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα ιδιαίτερα την οικονομική ανταγωνιστικότητα και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο στις εθνικές ανισορροπίες. Δεν πρέπει να τις τονίζουμε, αλλά να προωθήσουμε μία σύγκληση και θα πρέπει να φτάσουμε σε μία ισορροπία, εξισορρόπηση μεταξύ των περιφερειών, έτσι ώστε να προωθήσουμε συνολικά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να εξετάσουμε πτυχές διακυβέρνησης σε πολλά επίπεδα, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Και βεβαίως και η προσβασιμότητα από πλευράς των πολιτών έχει μεγάλη σημασία. Θέλετε να πείτε λίγα λόγια επειδή μου σε θίγησαν ενδιαφέροντα ζητήματα, δεν μπορούμε τώρα να αρχίσουμε μία συζήτηση. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά να γίνεται και άτυπα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί νομίζω ότι πολλά θέματα ήδη αναφέρθηκαν από διάφορους συναδέλφους. Εάν θέλουμε να θίξουμε το θέμα της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη σε, έναν, σε ένα παγκοσμιοποιημένο, παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Στην πολιτική συνοχή θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία των περιφερειών μας σε, αυτή την, σε αυτά τα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και πού, μάλλον σε ποιους τομείς πρέπει να εργαστούμε. Θα ήταν αντιπαραγωγικό να μιλάμε για παλαιά και νέα κράτη-μέλη, διότι η ανταγωνιστικότητα αφορά όλες τις περιφέρειες. Όταν μιλάμε για περιφερειακές, περιφερειακές ανισότητας, μιλάμε για ένα γενικότερο πλαίσιο, ορισμένες κοινές αρχές πολλές περιφέρειες ε, συγκλίνουν και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να θέσουμε επιτάπητος. Δηλαδή πώς μπορούμε να άρουμε τις διαφορές μέσα σε μία ίδια περιφέρεια και να ορίσουμε ε, ένα σύνδεσμο μεταξύ αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας και την όλη στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Χρειάζεται μια βιώσιμη ανταγωνιστικότητα η οποία να προσαρμόζεται σε θέματα κλιματικών αλλαγών, ε, ερήμωσης της υπαίθρου και να δούμε πώς ε, μπορεί να δράσει μια πραγματική πολιτική συνοχής. Ελπίζω ο συνάδελφος να συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε το μελλοντικό έγγραφο να μας εκφράζει όλους. Ο κύριος Λούχαν, σας παρακαλώ μην ασχοληθείτε με κάθε σημείο χωριστά. Σας ευχαριστώ από βάθους καρδίας διότι συνεισφέρατε στην όλη συζήτηση του θέματος της ε, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που είναι απαράβατος όρος ε, για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξ αρχής θα ήθελα να πω ότι δεν θα αναφερθώ στα 12 κράτη-μέλη που πιο πρόσφατα προσχώρησαν. Απλώς λέω ότι η κατάσταση είναι διαφορετική για τα 12 αυτά κράτη-μέλη όπως κατέδειξαν ορισμένες έρευνες. Αλλά δεν θα αναφερθώ μόνο στα 12 αυτά κράτη-μέλη. Είπα ότι θα πρέπει να εντάξουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο αυτό συνοχής. Αυτό είναι το καθήκον της έκθεσης. Τώρα, πώς θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Μία ιδέα ήταν η εξής. Να δούμε τις περιφερειακές ανισότητες. Αυτές ιδιαίτερα που είναι πολύ μεγάλες και οι ιδιαιτερότητες πολλές φορές είναι πολύ μεγάλες. Εδώ μιλώ για ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Πώς μπορούμε να ορίσουμε μία ενιαία συνεκτική δομή έτσι ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Και εδώ δεν μιλώ για παλαιά και νέα κράτη-μέλη. Χαίρομαι διότι το ανέφερε αυτό και ο συνάδελφος Ματούλα, διότι τόνισε το θέμα της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Ο κύριος Όλμπριχτ αναφέρθηκε σε ορισμένα στοιχεία ή μία κατονομασία της έκθεσης Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συγκεκριμένες επενδύσεις οι οποίες να είναι κατάλληλες για να αντιμετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών και εάν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις ιδιαιτερότητες δεν θα είμαστε συνολικά ανταγωνιστικοί. Θα σας αποστείλω ένα έγγραφο με mail για ένα προσχέδιο εγγράφου ή έκθεσης και μπορείτε να μου απαντήσετε σε οποιοδήποτε σκέλος θελήσετε. Ευχαριστούμε. Στις 26-27 θα ε, υποβληθεί έκθεση και η επόμενη έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με την χρηστή διακυβέρνηση. Θα ήθελα και εσείς να είσαστε, να είσαστε ιδιαίτερα σύντομος. Αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν με ακούει. Άρα μιλώ στον αέρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Έχετε μπροστά σα ένα έγγραφο εργασία το οποίο αναφέρεται στη χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στι διαδικασίε συνδρομή και ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έγγραφο λοιπόν εργασία έχει δύο τμήματα που άλλο συμπληρώνονται. Αναφέρουμε επίση τη Λευκή Βίβλο τη Επιτροπή των Περιφερειών που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2009. Όσον αφορά το πρώτο τμήμα του εγγράφου εργασίας, σε αυτό αναφέρομαι σε μία σειρά αξιολογήσεων και εκθέσεων και αναφέρομαι και σε κάποιες προτάσεις που κάνει η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής των Περιφερειών και έχοντας ως βάση την ανάλυση αυτή, λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν στην μελλοντική έκθεση τα ακόλουθα σημεία η σημασία που έχει η κάθετη και οριζόντια διάσταση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Είναι σημαντικό να έχουμε μία συνεργασία των εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών και να έχουμε όμως και μία συνεργασία μεταξύ παραγόντων του ιδίου επίπεδου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μόνο αυτό θα μπορούσε να εξασφαλίσει μία σφαιρική προσέγγιση ολοκληρωμένη σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη χρειάζεται μια, ένας καλύτερος ορισμός της εταιρικής σχέσης. Έχοντας ένα σαφέστερο ορισμό θα προχωρήσουμε σε καλύτερες, σε πραγματικές εταιρικέ σχέσεις, οι οποίες θεωρώ ότι δεν έχουν απτυχθεί όσο θα έπρεπε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ακόμα. και είναι πολύ σημαντικό να ενδυναμωθεί και η αρχή της διαβούλευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο προτού συζητηθούν κάποια ζητήματα σε κοινοτικό επίπεδο. Επίσης, πρέπει να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τις δυνατότητες που μας δίνει η εδαφική συνοχή και εδώ πέρα αναφέρομαι στην συμμετοχή των εθνικών και υπεθνικών παραγόντων στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέω ουσιαστικά ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε μια αποτελεσματική εφαρμογή της εδαφικής συνοχής. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε προδιαγραφές οι οποίες να τηρούνται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε καλύτερα την πολιτική συνοχής. Οι τελευταίες τροποποίησεις που γίνανε στον κανονισμό, ιδίως στον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μας βοήθησαν να ανταποκριθούμε καλύτερα στις νέες συνθήκες οι οποίες προέκυψαν. Επίσης, αναφέρομαι στο πρόγραμμα Εράσμους για τους τοπικούς και τους περιφερειακούς αντιπροσώπους. Για το σημείο αυτό λέω ότι θα πρέπει να δοθούν ε, οι απαραίτητοι πόροι, η απαραίτητη χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προσεχών διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό και λέω επίσης ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η δικτύωση με τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και στη συνέχεια αναφέρομαι στον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ένα τέτοιο έγγραφο που θα αναφερόταν στον χάρτη αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό μέσο για την ανάπτυξη μιας κοινή προσέγγισης της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Στο δεύτερο τμήμα του εγγράφου εργασίας αναφέρομαι στους ε, μηχανισμούς κοινή διαχείρισης. Και ειδικότερα αναφέρομαι στις διάφορες αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Και θα ήθελα να αναφερθώ εδώ πέρα στην ε, μεταφορά των αρμοδιοτήτων προς τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές προκειμένου να βελτιωθεί το σύστημα και πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και σχεδίων. Αναφέρουμε επίσης την ε, ενίσχυση την οποία μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ουσιαστικά τα περισσότερα ασφάλματα εντοπίζονται στο πρώτο επίπεδο ελέγχου. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα ελέγχου προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των ελέγχων. Αναφέρομαι επίσης στο εγγραφό μου στη συμμετοχή του ε, ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν καταφέρναμε να είχαμε κοινέ προδιαγραφές σε όλα τα σχέδια αυτά, η προσέγγιση θα ήταν πολύ καλύτερη. Σαφώς οι δικαιούχοι σε κάθε περίπτωση θα εποφεληθούν από τον συντονισμό των διαφόρων ταμείων και πόρων σε κοινοτικό επίπεδο. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας και εμεί στη θέση σας για οποιαδήποτε πρόταση έχετε να μου κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι μόλις τώρα ξεκινάει η συζήτηση για την ε, έκθεση αυτή. Θα έχουμε το σχέδιο έκθεσης πριν το καλοκαίρι. Ο Γιώργος Σταυρακάκης έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, μια που είμαι δίπλα σας. Θα προδίσω να σας ακούσω και θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έγγραφο εργασίας. Αποτελεί μια πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε και κάνει μια σωστή και εκτενή αναφορά πρώτον στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, οι οποίοι ως οι πλησιέστεροι στον πολίτη είναι και οι πλέον κατάλληλοι να παρέχουν πληροφορίες ή δεδομένα για τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο και δεύτερον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει το γενικό συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής. Μην ξεχνάμε αγαπητοί συνάδελφοι ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί ουσιαστικά τον χώρο όπου αναπτύχθηκε η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντική η αναφορά στην Λευκή Βίβλο της Επιτροπής των Περιφερειών για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας προγραμματικής περίοδου και στην αρχή της διαμόρφωσης της επόμενης, θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να προτείνουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για περαιτέρω βελτίωση του συστήματος πολιτικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής των Περιφερειών περιέχει αξιόλογες προτάσεις, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι θέτει πάρα πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες από τις προτάσεις της Λευκής Βίβλου μπορούν πραγματικά να υλοποιηθούν και να έχουν προστιθέμενη αξία για την περιφερειακή πολιτική και να εστιάσουμε αυτές. Πέρα από αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό με τις όποιες προτάσεις μας να καλύψουμε και τις πέντε αρχές στις οποίες εδράζεται η χρηστή κυβέρνηση. Δηλαδή, πρώτον, διαφάνεια, δεύτερον, συμμετοχή, τρίτον, ευθύνη, τέταρτον, αποτελεσματικότητα και πέμπτον, συνοχή. Τελειώνοντας, στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι μπορούμε να εξετάσουμε κάποιες περαιτέρω προτάσεις με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω της δέσμευσης των φορέων, όπως τη σύναψη τριμερών συμβάσεων, την conditionality ή το risk-based audit. Σας ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε, Όντσι Βιάσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Είμαι σαφώς υπέρ της α, ε, συνεχιζόμενης αυτής αποκέντρωσης, αλλά ας είμαστε σαφείς ως προς το εξής. Όταν αναφερόμαστε στους ε, κοινοτικούς σπόρους, θα πρέπει να, αγνο, να γνωρίζουμε ότι Ορισμένοι από τους σπόρους που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο εργασία έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιοχές όπως το Άμστερνταμ και το Ρότερνταμ. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι ε, το σύστημα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Το σύστημα ελέγχου είναι πάρα πολύ αυστηρό. Και οι θύνοντες στα διάφορα επίπεδα ουσιαστικά φοβούνται λόγω της μεγάλης ευθύνης την οποία φέρουν. Θα πρέπει λοιπόν όχι να αυξήσουμε τους ελέγχους, αλλά να απλοποιήσουμε την ομοθεσία, να απλουστεύσουμε την νομοθεσία ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν και νομίζω ότι ε, θα πρέπει επίσης να έχουμε και τα απαραίτητα προγράμματα κατάρτισης, είτε αυτό γίνει μέσω του Εράσμους, είτε μέσω ενός άλλου προγράμματος. Θα πρέπει οι τοπικοί και περιφερειακοί ηθήνοντες να λάβουν την απαραίτητη κατάρτιση προκειμένου να μην φοβούνται τις ευθύνες αυτές που έχουν στα πλαίσια της αρχής της ε, επικουρικότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μανέσκου για το εξαιρετικό έγγραφο εργασίας που σχετίζεται με θέματα χρηστής διακυβέρνησης σε πολλά επίπεδα. Μας ε, έδωσε ορισμένες ε, ιδέες σε σχέση με το ρόλο του ευρωβαρόμετρου και τις επιπτώσεις που υπάρχουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως δημοσιεύθηκαν στην έκθεση του 2009. Η έκθεση επιβεβαιώνει τις, ε, το, ε, επιθυμίες των ε, πολιτών και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα μέσω δημοτικών εκλογών βλέπουμε ότι το 59% των πολιτών θεωρούν ότι οι δημοτικές και τοπικές αρχές δεν λαμβάνονται υπόψη σοβαρά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό χαιρετίζω τις ε, ιδέες που υποβλήθηκαν θα πρέπει να έχουμε και οριζόντιες και εγκάρσιες σχέσεις εταιρικότητας για να φτάσουμε στο καταλληλότερο επίπεδο λήψης αποφάσεων όπου κυρίαρχο ρόλο θα παίζει ο πολίτης, ε, δηλαδή να μιλάμε για όλες τις διοικητικές υποδιαιρέσεις, φτάνοντας από τις τοπικές, τις ε, ε, δημοτικές αρχές, τις κοινοτικές και τις περιφερειακές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και τη διασυνοριακή συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και θα πρέπει να προωθήσουμε και την e-governance για να δούμε ποια είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις ε, αποφάσεις που λαμβάνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βίκτορ Βοστινάρου. Βίκτορ Βοστινάρου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, σε σχέση με αυτά που είπα στην προηγούμενη μου παρέμβαση, θα ήθελα να πω ότι είμαι υπέρ των βασικών ιδεών και της όλης φιλοσοφίας την οποία εισάγει σε αυτό το έγγραφο εργασίας η συνάδελφός μας κυρία Μανέσκου. Επίσης, θα πρέπει να εργαστούμε βάσει των ιδεών αυτών όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν και να σκεφτούμε δύο πράγματα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση των ιδεών αυτών. Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ισχύσει για τα κράτη-μέλη από την άλλη. Γιατί πέρυσι συζητήσαμε το ζήτημα της απλούστευσης αλλά η εφαρμογή του προγράμματος απλούστευσης σε ορισμένα κράτη-μέλη κατέστη πιο περίπλοκη, στα πλαίσια μάλιστα της απλούστευσης. Θα πρέπει λοιπόν και η απλούστευση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση να αποτελούν προϋποθέσεις, αν όχι για την υφιστάμενη πολιτική συνοχής, τότε για την πολιτική συνοχής που θα ισχύσει μετά το 2013. Αυτός θα πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος και για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την κυρία Μανέσκου για την έκθεσή της και θα ήθελα να της πω επίσης ότι εμείς θα συμβάλλουμε πάρα πολύ στην εξαιρετική αυτή έκθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μανέσκου, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και για τις συνεισφορές. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην ε, αποτελεσματικότητα της ε, χρήσης των ταμείων, έτσι ώστε να γίνεται σωστή χρήση τους από τους πολίτες μέσα στα πλαίσια ενός ελέγχου και εποπτείας, η οποία να ισχύει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και το ευεργέτημα να το καρπούνται οι πολίτες. Και όπως είπε και ο κύριος Σταυρακάκης, ε, αναφερόμενοι στις πέντε αυτές αρχές θα ακολουθήσω τις στοχοθετήσεις της στρατηγικής 2020. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη και ο Γιάνν Όλμπρικ ήθελε να πάρει το λόγο. Δεν σας είδα. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Δύο προτάσεις θα ήθελα να κάνω. Πιστεύω ότι εν γέννη το περιεχόμενο του εγγράφου εργασία είναι πολύ καλό, εύστοχο, αλλά θα μπορούσα να προτείνω το εξή. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε ότι ε, η όλη έννοια της εδαφικής συνοχής δεν χρησιμεύει σε τίποτα αν δεν έχουμε πολυπίπεδη διακυβέρνηση. Νομίζω ότι ε, είναι απόλυτα λογικό αυτό. Η εδαφική συνοχή τι σημαίνει ουσιαστικά. Ισορροπία ανάμεσα στις ε, διαφορετικές περιφέρειες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν ε, κάποιες περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν ε, προβλήματα. Από την άλλη μπορεί να έχουμε περιφέρειες οι οποίες είναι πιο σύγχρονες, πιο μοντέρνες, άλλες περιφέρειες πιο μικρές, άλλες περιφέρειες είναι μεγαλύτερες. Επομένως χρειαζόμαστε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στα πλαίσια της εδαφικής συνοχής και η συνεργασία αποτελεί πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και θα πρέπει να δείξουμε ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν είναι απλώς μία επιλογή ανάμεσα σε άλλες αλλά εκ των ουκάνευ προκειμένου να έχουμε μία πολιτική εδαφική συνοχής ότι επίσης υπάρχουν διάφορα εμπόδια, μπορούμε να πούμε ότι βάσει της αρχής της επικουρικότητας θα πρέπει αυτή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση να γίνει υποχρεωτική. Γιατί αν αφήσουμε την απόφαση αυτή στα κράτη-μέλη, ουδέποτε πρόκειται να ληφθεί ω δεσμευτική απόφαση. Νομίζω λοιπόν ότι στη μελλοντική έκθεση θα πρέπει να λέγεται ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι απολύτω υποχρεωτική και ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στην, στο σχέδιο έκθεση της κυρίας Κράτσα και θα έχουμε πάλι την 24η Μαρτίου στις 6 το απόγευμα προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Η κυρία Κράτσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα της έκθεσης έχει να κάνει με τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της χρηματοοικονομικής κρίσης με ιδιαίτερη αναφορά στο στόχο 2. Ε, στο έγγραφο που σας έχει ήδη κατατεθεί, στο σχέδιο έκθεση που έχει ήδη κατατεθεί, ε, ξεκινάω τονίζοντας τη σημασία που έχει η πολιτική συνοχής ε, για την ε, ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, όχι μόνο διότι είναι ένα δεδοκιμασμένο μέσον, αλλά διότι η, όπως αποδεικνύεται η έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών ε, οικονομικού και δημοσιονομικού συντονισμού και ισόρροπης ανάπτυξης στην Ευρώπη δίνει την, ε, ε, την έμφαση πια στην πολιτική συνοχή μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων εργαλείων να παίξει τον πρωταρχικό ρόλο που έχουμε ανάγκη για την ισορροπία της εσωτερικής αγοράς και της σύγκλησης. Υπενθυμίζω επίσης ότι η περιφερειακή πολιτική δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο άμεσης κατάσβεσης σε ε, εποχές κρίσης, που και εκεί είδαμε την ανθεκτικότητά της και την δημιουργικότητά της πολιτικής, αλλά είναι βασικά ένα ε, εργαλείο για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμα αδυναμιών των περιοχών. Και την εποχή της χρηματοοικονομικής κρίσης είδαμε και ανάδειξη ανάδυση αυτών των αδυναμιών όπως συμβαίνει πάντα στις κρίσεις που βγάζουν στην επιφάνεια τις αδυναμίες. Ε, επισημαίνω ότι ο στόχος 2 αποτελεί ε, ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες της πολιτικής συνοχής ε, και επειδή ακριβώς αναφέρεται στην ανταγωνιστικότητα αφενός και στην απασχόληση ε, πρέπει, ε, ε, αυτό είναι και το νόημα της έκθεσης πρωτοβουλίας, να δούμε την, τα αποτελέσματά του και την, να ενισχύσουμε το ρόλο του στην πολιτική μας για την έξοδο από την κρίση. κάνω μια αναφορά στο παρελθόν, υπεθυμίζοντας ότι στην περίοδο 2000-2006 ο στόχος 2 αφορούσε την υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης περιοχών που εμφάνιζαν αδυναμίες ιδιαίτερες διαρθρωτικές και <clears throat> εποφελήθηκαν ήδη ε, το 15,2% των Ευρωπαίων α, που ζούσαν στις περιοχές ε, το στόχου 2, ε, ενώ με τη μεταρρύθμιση του, ε, του 2006 ε, ο στόχος 2 αφορά την πλειονότητα των περιοχών και ο, επίσης ένα σημαντικό ποσό του συνολικού προϋπολογισμού περίπου το 16% των συνολικών πόρων και εστιάζεται ιδιαίτερα στην ανταγωνιστικότητα και στην ε, ε, απασχόληση. Ε, σημειώνω ότι το 73,7 περίπου του ποσού αυτού που αντιστοιχεί στο στόχο 2 προορίζεται για τη βελτίωση της γνώσης και της καινοτομίας, ε, είναι το ποσοστό του 33 περίπου της για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, περίπου το 40%, το αντίστοιχο ποσό για τις περιφέρειες του στόχου 1 είναι αισθητά χαμηλότερο, μόλις 40%, αν και σε απόλυτους αριθμούς υπερέχει σημαντικά λόγω των αυξημένων αναγκών των ε, ε, λόγω περιοχών. Ε, θέλω να πω με αυτά τα στοιχεία ότι προσανατολίζει το στόχος 2 σε τομείς εχμής όπως είναι η έρευνα, η καινοτομία, η ποιότητα των θέσεων εργασίας, στοιχεία ακριβώς που τα χρειαζόμαστε για την ανταγωνιστικότητα. Ε, βάσει τώρα τα, της τελευταίας έκθεσης πρόοδου Επιτροπής σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή, οι περισσότεροι δείκτες της περιφέρειας του στόχου 2, 2 σημείωναν πριν από την οικονομική κρίση υψηλέ επιδόσεις, όπως την απασχόληση, την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη, την ένταση ε, ανθρωπίνου δυναμικού, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, τη διαβίου εκπαίδευση, ε, ενώ σε άλλους όπως η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων ε, και της παραγωγικότητας, οι περιφέρειες σύγκλησης σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις. Ε, λόγω του ότι εκεί υπάρχει ανάγκη για άλλη κατεύθυνση ανάπτυξης, για βασικές ε, επενδύσεις. τονίζω, δίνω αυτά τα στοιχεία αντιπαραβάλλω για να δείξω ότι είναι, έχει κατεύθυνση στην ποιότητα και στην ανταγωνιστικότητα και το οποίο είναι ήδη σαφές από τα αποτελέσματα. Ε, ε, τώρα που η οικονομική κρίση αναδεικνύει, ε, όπως είπαμε, όχι μόνο τις αδυναμίες των περιοχών, αλλά και τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής σύγκλησης προς την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση των ευρωπαϊκών περιοχών, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προβλέψεις για το 2009-2011 της Επιτροπής, ε, σύμφωνα με τις οποίες η κατάσταση της αγοράς εργασίας θα παραμείνει δυσμενής, το ποσοστό της ε, ανεργίας προβλέπεται να ανέλθει στο 10,25% με απώλεια του 2,25% των θέσεων εργασίας για το 9 και κάτι παραπάνω από το 1% για το 2010. Ήδη λοιπόν ε, έχουμε τα πρώτα δείγματα της ανάγκης αξιοποίησης και εντατικοποίησης των προσπαθειών ε, για τις περιοχές ε, του στόχου 2. Ε, ήθελα να ε, επισημαίνω επίσης βέβαια και τους τομείς στους οποίους αναφέρομαι και στους τομείς στους οποίους υπάρχουν τα αποτελέσματα και οι προβλέψεις για την, για την επίδραση του, των πολιτικών μας του στόχου 2 ε, και όμως ε, ε, επισημαίνω ότι τα μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα πολλών κρατών αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα και τροχοπέδι στη συμβολή εθνικών συγχρηματοδοτήσεων στα προγράμματα που αφορούν το στόχο 2. Είναι κάτι δεδομένο και ισχύει για όλες τις χώρες. αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη ε, από στοιχεία συγκεντρωτικά, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά για τις ε, ε, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης ε, και στη διαμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών δικτών και γι' αυτό για να μπορέσουμε να είμαστε πιο σαφεί στην παρέμβασή μας και στις συστάσεις μας και στις κατευθύνσεις που θα ζητήσουμε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια ειδική έκθεση για τις συνέπειες της κρίσης στις περιοχές του στόχου 2 με δεδομένο αυτές τις προβλέψεις και τη, ήδη αποτελέσματα που έχουμε επισημάνει. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να γίνει ένα συντονισμό και κινητοποίηση όλων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μα. Όπω συζητήσαμε και στην πρώτη παρουσίαση του θέματο, ε, υπάρχουν ε, πολλά ε, μέσα τα οποία δρούν στην, για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και θα πρέπει να γίνει ένα συντονισμό όλων αυτών των μέσων για, για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και μακροπρόθεσμης παρέμβασης για τις αδυναμίες. Ε, ήδη το θέμα τονίστηκε ιδιαίτερα και τονίζεται και στην έκθεσή μου το θέμα των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων που πρέπει να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες της ε, διευκόλυνσης χρηματοοικονομικής αλλά και των επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία. Ήδη είδαμε τα προβλήματα που ήδη έχουν, συγκεντρώνονται ως επιπτώσεις της κρίσης στην πραγματική οικονομία ε, και ε, τις δυσκολίες λόγω του ότι ε, σε αρκετές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις διάσωσης μπορεί να είναι δυνητικά ασύμβατες με τις πολιτικές για τον σωστό ανταγωνισμό. Γι' αυτό πρέπει να γίνει η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που βοηθούν ουσιαστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν έχουν ανάγκη μόνο την άμεση ενίσχυση για τη διάσωσή τους. Ε, κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει οι προβλέψεις μας να ενταχθούν μέσα στο μακροπρόθεσμο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατηγική 2020 ε, και να συνδεθεί με την κοινωνική και την εδαφική συνοχή της Ένωσης, διότι η, η, ο στόχος της ανταγωνιστικότητας έχει να κάνει και με το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η προσπάθεια για εδαφική συνοχή. Ε, και αναφέρομαι ιδιαίτερα, δεν τονίζεται αλλά εννοείται, ε, οι νησιωτικές ε, περιοχές, οι αποκεντρωμένες περιοχές, διότι και αυτές έχουν μερίδιο στον αγώνα για την ανταγωνιστικότητα. Επίσης, η προσπάθεια για αηφόρο ανάπτυξη, για πράσινο ανάπτυξη, δίνει και αυτή μία δυνατότητα στις, στην προώθηση των πολιτικών για το στόχο 2. Ε, παράλληλα, πρέπει να εφαρμόσουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο όλες τις απλουστεύσεις που δόθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης, ε, που έχουν να κάνουν με νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα ε, για τη μεγαλύτερη ελαστικότητα στα προγράμματα συνοχής, την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των περιφερειών σε αυτές τις διευκολύνσεις, ε, και φυσικά την κατεύθυνση και την υποστήριξη για τις έξυπνες ε, επενδύσεις. Ε, βλέπουμε από τις πρώτες εκθέσεις, τις εθνικές εκθέσεις που έχουν καταθέσει τα κράτη-μέλη ότι δεν έγινε παντού η ίδια αξιοποίηση αυτών των διευκολύσεων. Πολλά κράτη-μέλη είχαν συνηθίσει σε ένα ρυθμό γραφειοκρατικό, διοικητικό και δεν έκαναν την αξιοποίηση αυτών των μέσων. Παραδείγματο χάρη την ε, προχρηματοδότηση του 100% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε, ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει πιο συστηματικά να, να δούμε πώς θα γίνει η χρήση αυτών των διευκολύνσεων ε, για την, που έχουν σχέση με την ελαστική και παράλληλα συνεπή ε, ε, εφαρμογή των ε, κανόνων και των ελέγχων, διότι από τη μια μεριά πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι και πιο αποτελεσματικοί, από την άλλη μεριά όλο περισσότερο πιο διαφανής και συνετή στη διαχείριση. Και ήθελα επίσης να τονίσω για την πολιτική βοήθεια για τα μεγάλα σχέδια για τις περιφέρειες του στόχου 2 που σήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έπαιξε θετικό ρόλο. Πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω την αύξηση άνω του 25% των παρεχομένων χρηματοδοτήσεων μέσω του Jaspers ε, με στόχο την προετοιμασία και τη γρήγορη εφαρμογή των μεγάλων σχεδίων και την επιτάχυση των πληρωμών στα κράτη-μέλη ε, και πρέπει επίσης ε, να υποστηρίξουμε και όλους τους άλλες αλλαγές, τους εκτελεστικούς κανόνες που επιδιώκουν να ενισχύσουν αυτή την ε, ευελιξία. Είχαμε κάνει και μια συζήτηση σχετικά με τον πρόεδρο της ε, ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, διότι επαναλαμβάνω κλείνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που δίνονται αφενός για τα μεγάλα σχέδια. Η ανταγωνιστικότητα χωρίς μεγάλα σχέδια δεν μπορεί να επιδιωχθεί και από την άλλη πλευρά η πρόσβαση σε διευκολύσεις των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, αυτό λοιπόν έτσι είναι και ένα τελικό μου μήνυμα. Ε, η σημασία της, της πολιτικής συνοχής, ιδίως μέσα στο πλαίσιο των αδυναμιών που ανέδειξε στην εσωτερική μας αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η, η, κρίση και δεύτερον η κινητοποίηση και ο συντονισμός όλων των εργαλείων που διαθέτουμε την επίτευξη αυτού του στόχου και η αξιοποίηση των ο, η αξιολόγηση και αξιοποίηση των μέτρων που ήδη τέθηκαν σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση της κρίσης θα, είναι, ε, θα μπορούμε να εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα όταν θα έχουμε ε, την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Εθνικών ε, Reports. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βεστφάλη είναι η πρώτη που έχει πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ακούσαμε η Οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιπτώσει σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις ε, στην Ευρώπη, όχι μόνο στα πιο φτωχά κράτη, αλλά ιδιαίτερα στις περιφέρειες, ε, περιοχής του στόχου 2. Η έκθεση κυρία Κράτσα είναι μια πολύ καλή συμβολή. Τονίζει δικαίως ότι στους ε, περιφέρειες στόχου 2 δημιουργήθηκαν 720.000 θέσεις απασχόλησης με 22 δισεκατομμύρια ενίσχυση. 314.000 ε, άνθρωποι στην Ευρώπη ωφελήθηκαν από την περιφερειακή ενίσχυση. Κατά τη γνώμη θα πρέπει όμως η έκθεση να τονίζει περισσότερο τις κοινωνικές ε, πτυχές της καταπολέμησης της κρίσης. Για μας τους Ισουροδημοκράτες οι εργαζόμενοι είναι στο επίκεντρο της καταπολέμησης της κρίσης. Θέλουμε και πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε κατά περισσότερες θέσεις απασχόλησης και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης εκεί που αυτές έχουν χαθεί. Αυτό ο τομέας θα πρέπει να ληφθεί περισσότερη υπόψη στην ελόγω έκθεση. Από σκοπιάς μας, οι προτεραιότητες της στρατηγικής για το 2020 που αναφέρονται στο σημείο 4 της έκθεσης δεν είναι επαρκής. Ανταγωνιστικότητα, ενίσχυση των επιχειρήσεων, ανάπτυξη των ΜΜΕ. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά δεν αρκούν. Θέλουμε να έχουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και καλύτερους όρους εργασίας. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε όμως και καλύτερες δυνατότητες εκπαίδευσης και μεταεκπαίδευσης, όχι μόνο για τους νέους, αλλά ιδιαίτερα για τους νέους. Παράδειγμα, ε, ίδιο μισθό για την ίδια εργασία για άντρε και γυναίκες σε όλη την Ευρώπη. Ξέρουμε ότι σε μια χρηματοπιστωτική κρίση οι γυναίκες είναι εκείνε που υποφέρουν ιδιαίτερα και που πρώτες χάνουν τη θέση εργασίας τους. Οι γυναίκες ιδιαίτερα γιατί θεωρείται ότι απλώς εκείνες προσθέτουν στο οικογενειακό εισόδημα ή επειδή έχουν τις χειρότερες θέσει εργασία. Είναι σαφέ. Οι επιπτώσει τη χρηματοπιστωτική κρίση στην οικονομία δεν θα πρέπει να ε, μας κάνουν να παραβλέπουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και καλύτερη κατάρτιση. Το σημείο 12 της κύριε Κράτσα μου φαίνεται ότι είναι προβληματικό. Η αύξηση των πόρων για το πρόγραμμα Jasper. Θα πρέπει καταρχήν να δούμε η αύξηση των κονδυλίων που προέβλεψε η Κομισιόν το 2009 κατά 25% πώς χρησιμοποιούνται και ποια είναι τα αποτελέσματά του πριν ζητάμε περισσότερα χρήματα. Και ήρθε εδώ το ερώτημα, από πού θα προέρχονται τα χρήματα αυτά και γιατί θα χρησιμοποιούν τα εν λόγω κονδύλια στην διοίκηση ή σε πραγματικά σχέδια. Εκτός αυτού, οι για το 2010 αυξήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από 24 σε 26 εκατομμύρια. Και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται περισσότερη αύξηση χωρίς να διευκρινιστούν τα ερωτήματα που σας παρουσίασα. Γενικά όμως εμείς οι σοσιαλδημοκράτες θεωρούμε ότι η έκθεση είναι το σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει και στο μέλλον να τομινίζεται ιδιαίτερα στις περιφέρειες του στόχου 2. 314 εκατομμύρια Ευρωπαίων θα μας είναι ευγνώμονες. Sí, gracias, Presidenta. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κράτσα για την έκθεσή της. Γνωρίζουμε ότι η πολιτική συνοχής δεν αφορά μόνο υποστήριξη από τον προϋπολογισμό, δηλαδή δημοσιονομική υποστήριξη, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε τις περιφερειακές δαπάνες, ιδιαίτερα του στόχου 2. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ρόλο των ΜΜΕ καθώς και των κέντρων καινοτομίας. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες μπορούν να προβλέψουν τις ανάγκες των ΜΜΕ και των εργαζομένων. Ο, οι περιφέρειες του στόχου 2 ε, καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης ε, μέτρων για την αντιμετώπιση της ε, κρίσης, για την ανάπτυξη και την οικονομική συνοχή. Ευχαριστώ. Ε, ένα θέμα θα ήθελα να ε, αναφέρω μπορείτε να μας πείτε πώς έχει το χρονοδιάγραμμα διότι είναι πολύ καλή η έκθεση, είναι πολύ δυνατή η έκθεση ως προς τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές που θα πρέπει να προβάλλουμε για μια ανάκαμψη. Έχουμε και την Επιτροπή Αντιμετώπισης της Κρίσης. Δεν ε, άκουσα τίποτα για τη δράση αυτής της Επιτροπής, αλλά θα πρέπει εμείς να μπορέσουμε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ε, ώστε να συνδράμουμε ως προς το σκέλος της πολιτικής συνοχής. Νομίζω ότι θα πρέπει να εισακουστεί αυτή η έκθεση. Ίσως μπορεί η συγγήτρια να μου δώσει ορισμένες πληροφορίες ως προς το χρονοδιάγραμμα, διότι δεν πρέπει να σταματήσει εδώ η έκθεση αυτή. Θα πρέπει να κινηθεί και προς αλλού. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, κύριε Στόιρερ, ω ε, σκιοδοσηγητή για την ε, ομάδα Άλτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια για την τόσο καλή έκθεσή της που αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τη συζήτηση του τόσο σημαντικού θέματος. βάνει πολλά θέματα, σημεία με τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν ίσω κάποια σημεία που κατά τη γνώμη μου ε, θα πρέπει να συζητηθούν ή και να τροποποιηθούν. Γενικά όμως όσον αφορά το στόχο 2 θεωρούμε μέσα στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης βλέπουμε να υπάρχει μια μετατόπιση ή ίσως μια επανεκτίμηση του στόχου αυτού γιατί όπως λέτε και στην πρώτη αιτιολογική σκέψη η απόσταση μεταξύ των περιοχών ε, στόχου 1 και στόχου 2 έχει μειωθεί. Καταρχήν επειδή υπήρχε μια επιτυχής ε, πολιτική για τις περιφέρειες ε, στόχου 1 και επειδή στο στόχο 2 υπήρχε επιδείνωση της κατάστασης. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την... σε εξελίξη του 2008-2009 όπου έχουμε ένα μείον 8, 10, 12% Και νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η κοινωνική συνοχή δεν σημαίνει ότι πιο αδυν, δυνατοί θα πρέπει να γίνουν πιο αδύναμοι, των αντίων οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να γίνουν πιο δυνατοί. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα περάσουμε στο τομέα της ανάπτυξης πάλι. Δηλαδή τώρα που δίθεται το θέμα της αξιολόγησης των διαφόρων στόχων θα πρέπει εδώ να πω ότι τα μέτρα της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να εστιαστούν στην ανάπτυξη, όχι στην διατήρηση δηλαδή κάποιας δομής, αλλά στην προσαρμογή των δομών, και καινοτομία, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Και ακριβώς ε, η περιφερειακή ενίσχυση στον τομέα του στόχου 2 πολλά μπορεί να προσθέσει εδώ, να προσφέρει και αυτό αναφέρεται και ξεκάθαρα στην έκθεση. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το θέμα της μεταφοράς της τεχνολογίας, δηλαδή οι γνώσεις να περνάνε από τις, τα ερευνητικά κέντρα στις επιχειρήσεις με την ανάπτυξη νέων προϊόντων που μόνο τα νέα προϊόντα μπορούν να δημιουργήσουν ε, σταθερές θέσεις απασχόλησης. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πτυχή του περιβάλλοντος. Γιατί πραγματικά η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί με τεχνολογική ανάπτυξη. Η τεχνολογική ανάπτυξη είναι και η βάση για την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα πρόβλημα έχουμε και δεν θα μακρηγορήσω περαιτέρω. Έχουμε λέω με την προχρηματοδότηση με το λεγόμενο front loading δεν με ικανοποιεί αυτό που προτείνεται αυτή τη στιγμή, γιατί θα πρέπει να διακρίνουμε με το ξύ του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου για την Περιφερική Ανάπτυξη και ξέρω ότι και αυτή είναι και η άποψη στο Συμβούλιο ότι υπάρχουν καλοί λόγοι για την συγχρηματοδότηση. Συγχρηματοδότηση σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στα σχέδια έχουν κάθε συμφέρον τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν σωστά. Ε, είναι θέμα δηλαδή αποτελεσματικότητας. Όχι απλώς να τρέχουμε πέρα εδώ θα να επιτυχάνουμε τίποτα, αλλά να προβλέπετε κάτι που τελικά καρποφορεί και εδώ νομίζω ε, μια ίδια συμβολή είναι ένα καλό μέσο. Ίσως θα μειώσουμε το ποσοστό, αλλά να το διαγράψουμε τελείως μου φαίνεται υπερβολικό. 100% ε, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προβληματικό κατά τη γνώμη μου και γενικά θα πρέπει να υπάρχει συγχρηματοδότηση. Έτσι βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα πράγματα σίγουρα και θα υποβάλουμε και μια σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λέει η κυρία Ντέλη, σας ζητώ συγγνώμη μου να στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Διάβασα όμως πολύ προσεκτικά την έκθεση και θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια του στόχου 2 να επενθυμίσουμε την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος και ότι θα πρέπει στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων να μπει και η διάσταση της βιωσιμότητας. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφαιρθούμε στον σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις για τον στόχο 2. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πολύ μεγάλη σημασία πλέον στην ε, αστική διάσταση όσον αφορά την εδαφική συνοχή και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στην ε, έκθεση αυτή να γίνεται αναφορά στο ότι οι, οι περιφέρειες του στόχου 2 θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στο ζήτημα των πόλεων και κυρίως των περιοχών εκείνων που είναι υποβαθμισμένες. Επίσης θεωρώ ότι το κείμενο αναφέρεται επιλεκτικά σε κάποιες προτεραιότητες στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αναφέρεται στην πολύ σημαντική προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην αηφόρο ανάπτυξη και στην καλύτερη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να καταφέρουμε να περάσουμε σε μια οικονομία που θα χρησιμοποιεί περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πηγές ενέργειας οι οποίες εκπέμπουν χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Το κείμενο επίσης δεν αναφέρεται ρητός στην ε, προτεραιότητα της ε, αποκλειστικής ε, ανάπτυξης. Ένα τμήμα της στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα. Μία από τις προτεραιότητες με την οποία όλοι συμφωνούμε είναι να συνεχιστούν οι στόχοι της πολιτικής κοινωνικής συνοχής. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να επανοριστούν οι δείκτες που θα μας επέτρεπαν να αξιολογήσουμε την κρίση χρησιμοποιούμε μέχρι στιγμής τα κλασικά όργανα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας όπως η οικονομική ανάπτυξη και το ΑΕΠ. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν και άλλα κριτήρια και άλλοι δείκτες προκειμένου να κάνουμε την αξιολόγηση αυτή. Η στρατηγική της Λισαβόνας είχε επικεντρωθεί πάρα πολύ στην ανταγωνιστικότητα Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, αν θέλετε, την κρίση αυτή, προκειμένου να υιοθετήσουμε μια νέα, μια νέα προσέγγιση και να εξασφαλίσουμε την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ο Μπρούνο Κασέτ, εξ νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλει να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον το οποίο δείχνει για την συνέχιση των μέτρων που έχουν ληφθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση και οι ε, επιπτώσεις κρίσης αυτής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια της ζήτησης αυτής θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτον, στα πλαίσια των ε, μέτρων παρακολούθησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να ξεκινήσει μία μελέτη για τις ε, ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις της κρίσης ε, όσον αφορά τα βασικά λειτουργικά προγράμματα της πολιτικής συνοχής και κατά αυτόν τον τρόπο απαντούμε επίσης και στη σχετική ανησυχία της εισηγήτριας κυρίας Κράτσα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το καλοκαίρι θα υποβάλει μία έκθεση για την χρησιμοποίηση όλων των μέσων της πολιτικής οικονομικής ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή διάσταση για όλα τα κράτη-μέλη και σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως αυτές παρουσιάστηκαν την 1η Απριλίου του 2009. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, θα ήθελα να ζητήσω από τη Ρόδη Κράτσα να μας πει αν θέλει να απαντήσει σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Φυσικά θα ήθελα να απαντήσω και να ευχαριστήσω καταρχάς τους συναδέλφους για τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις που έκαναν. Φαίνεται από αυτό ότι το θέμα μας απασχολεί όλους και το θεωρούμε δομικό για τα επόμενά μας βήματα. Ε, ήθελα καταρχάς να μείνω με προσοχή στις κοινωνικές επιπτώσεις. Είναι και στη δικό μου σκεπτικό με κάποια τροπολογία να ενισχύσω τον τομέα αυτό, διότι αφαίρεσα αρκετά πράγματα από όσα είχα σκοπό να εισάγω λόγω του, ξέρετε, του άγχους του περιορισμού του, της έκτασης. Ε, για τις γυναίκες, παρόλο που είναι ένα θέμα που το αγαπώ και το υπηρετώ ιδιαίτερα, δεν είχα σκοπό να παρέμβω, διότι τα προβλήματα αυτά της αντιμετώπισης των διακρίσεων, της σημασίας τους για την κοινωνία της συνοχής, έχουν τη θέση τους σε πολλές ε, άλλες ε, ευκαιρίες, εκθέσεις, ψηφίσματα ε, και εξάλλου το θεωρώ ότι είναι κάτι δεδομένο σαν όρος αξία και στόχος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Για το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ε, αναπόφευκτο ε, συζητήθηκε και με την αφορμή προηγούμενων, παρουσίας προηγούμενων εκθέσεων ότι χωρίς ε, τις τοπικές περιφερειακές αρχές που έχουν την ευθύνη της εφαρμογής, της τελικής εφαρμογής των πολιτικών μας δεν μπορούμε να επιδιώξουμε τους στόχους μας. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω, θεωρώ πολύ σημαντικό, το, την ένταξη της αστικής διάστασης ε, η πόλη είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την ανταγωνιστικότητα. Συνήθως είναι οι αιστείες της καινοτομίας, της ανάπτυξης, η πόλης, αλλά εκεί συσσωρεύονται και τα περισσότερα κοινωνικά προβλήματα και θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την αστική διάσταση, όπως και για την ε, αηφόρο ανάπτυξη. Ε, και το άλλο που ήθελα να απαντήσω ιδιαίτερα είναι για το 100% της προχρηματοδότησης. Ε, ε, θεωρώ ότι λογικά όταν υπάρχει συγχρηματοδότηση υπάρχει και συνυπευθυνότητα, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε σε ένα τέτοιο πλαίσιο σήμερα όπου μια διευκόλυνση ε, σε μια εποχή κρίσης, σε μια εποχή δυσκολίας δημοσιονομικής που έχουν τα κράτη-μέλη, μπορεί να μας βγάλει έξω από το πλαίσιο της συνυπευθυνότητας αφού οι κανόνες είναι εκεί και στο τέλος θα δοθεί οπωσδήποτε ο λογαριασμός. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι μια πρόταση, δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί και ήδη πολλές χώρες δεν το έχουν αξιοποιήσει αυτή τη διευκόλυνση του 100%. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελέτη, που θα, που, τη μελέτη των επιπτώσεων που ετοιμάζει, αλλά και την αξιοποίηση των εργαλείων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων πράγματι απαντά σε μια ανησυχία της ε, έκθεσης και σε ένα συγκεκριμένο αίτημα. Και όσο για τις προβλέψεις ε, που ζήτησε ο κύριος Νιστερό, ήθελα να πω ότι η βασική μας πρόβλεψη ήταν να υιοθετηθεί τον Απρίλιο η έκθεση. Αν ε, η Επιτροπή μας πιστεύει ότι πρέπει να αναμένουμε άλλες εξελίξεις και να την υιοθετήσουμε αργότερα, εγώ είμαι στη διάθεσή σας να ακολουθήσουμε τον ρου του Κοινοβουλίου είναι ότι νομίζετε ότι είναι το καλύτερο για να μπορέσει να αποτυπώσει πράγματι ε, το κεκτημένο και τις αποφάσεις ε, που, από θέματα που επεξεργάζονται ήδη σε άλλες ε, επιτροπές. Σας ευχαριστώ πολύ. I, I thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, γιατί ίσως υπήρχε κάποιο παρεξήγηση. Το ο κύριος Φανίστερόι, από ό,τι κατάλαβα, είπε ότι θα πρέπει να εργαστούμε πάνω σε κάτι που θα μπορεί να συμβάλλει στη συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή για την κρίση. Και εγώ θέλω να σας πω ότι σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατάφερα μέσω της εθνικής μου να περάσω σαν ε, ε, συμπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Κρίσης. Και έχω να πω ότι υπάρχει και η κρίση αυτή στην πραγματική οικονομία και αυτό είναι κάτι που πλήττει όχι μόνο το εθνικό επίπεδο αλλά και πολύ ανά το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και υπάρχει και η πολιτική συνοχή που τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε μια συμβολή στην ε, ε, πολιτική, πολιτική καταπολέμηση της κρίσης και έχουμε μία έκθεση η οποία θα συμβάλλει στην κύρια έκθεση για την ε, κρίση. Η κύρια έκθεση προετοιμάζεται από την κυρία Περβάν Περές και η δική μου συμπληρωματική έκθεση είναι ακριβώς για τη συμβολή της ε, πολιτικής συνοχής στην ανάκαμψη και σε σχετισμό με τη μακροπρόθεσμη ε, ανάκαμψη και αν η κυρία Κράτσα ολοκληρώσει την εκθεσή στον Απρίλη θα συμβάλλει και αυτό πάρα πολύ στη συζήτηση για την ε, κρίση και για την καταπολέμηση της κρίσης και τις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Το κύριο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τις επιπτώσεις της κρίσης στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα, στικά, τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι και πολύ συγκρίσιμα και δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά. Θα τα έχουμε πολύ αργότερα. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε εθνικά στοιχεία για την κρίση από ότι περιφερειακά και τοπικά. Έγιναν όμως διάφορες παρατηρήσεις από ενώσεις περιφερειών που συμβάλλουν ε, στην κατανόησή μας για τις επιπτώσεις αυτής της ε, κρίσης σε, εθνικό, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι μια συμπληρωματική παρατήρηση μονάχα. Α, με συγχωρείτε κυρία Γράτσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την ε, πρόταση συνεργασίας και αξιοποίησης της δουλειάς που κάνουμε εδώ στο πλαίσιο της ε, ε, γενικότερης προσέγγισης της απάντησης στη δημοσιονομική κρίση που επεξεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να απαντήσω για το θέμα των μεγάλων έργων, της αύξησης αυτό στα μεγάλα έργα. Είναι κάτι που εγώ το υποστηρίζω. Δεν μπορεί να επιδιώκουμε ανταγωνιστικότητα χωρίς την διευκόλυνση της προετοιμασίας για τα μεγάλα έργα. Εξάλλου δεν είναι τόσα πολλά αυτά που γίνονται στα, στο στόχο 2, είναι τα περισσότερα στις ε, περιοχές σύγκλησης και πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία την εποχή που ε, περιορίζονται οι δημόσιες δαπάνες από τα κράτη-μέλη λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών, να υπάρχει διευκόλυνση οραματισμού και προετοιμασίας μεγάλων έργων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμένη μου πολύ τροπολογίων, όπως σας είπα, είναι 24 Μαρτίου στις 6 το βράδυ. Προθεσμία για τις τροπολογίες 24 ε, Μαρτίου 6 το βράδυ. Τώρα έχουμε μερικά λεπτά για το σημείο 10 που όπως θυμάσαστε το αντικαταστήσαμε το σημείο 7 με το σημείο 10. Μια σύντομη παρουσίαση για τη συνεδρία της ομάδας εργασίας σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή. Είχαμε τη δεύτερη συνάντηση και παραδοσιακά καλούμε τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο, για να παρουσιάσει την τρέχουσα εργασία για το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή. Για μετά το 2013 και ακούσαμε τον κύριο Νίκολα Ντεμικελής που τώρα είναι επικεφαλής του γραφείου του νέου Επιτρόπου Γιώχανες Χάν και ο Έρικ Βαμπρέσκα που είναι ε, σε στο, στη στο τμήμα που αφορά και ασχολείται με τα θέματα αυτά της μελλοντική πολιτικής. Ε, Συστήσαμε πολλά θέματα στο παρελθόν όσον αφορά τη μελλοντική μορφή και στόχους της πολιτικής συνοχής και την απλούστευση του συστήματος. και συνοχή, υπήρχε μια ανεπίσημη ανταλλαγή απόψε να προς το τέλος της συνεδρίασης. Συμφωνήσαμε στην ακολουθητέα διαδικασία, γιατί είπαμε ότι για να υπάρχουν επιπτώσεις ε, της ε, πολιτικής αυτής, θα πρέπει εμείς κάτι να παρουσιάσουμε σαν Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Και είναι καλό να έχουμε κάποιον επίσημο έγγραφο ίσως, με ορισμένα βασικά πολιτικά στοιχεία. Που θα μπορούσε η ομάδα εργασία να τα υιοθετήσει, ας πούμε, σαν πρόταση να προωθηθεί και να επικυρωθεί στις συνεδρίες του Ιουλίου ίσως, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στην Κομισιόν αυτό το σημείο, τους βασικούς όρους δηλαδή, καθημάς της μελλοντική πολιτικής συνοχής. Χωρίς να μπούμε στις λεπτομέρειες, αλλά τουλάχιστον για να έχουμε ένα σημείο εκκίνησης. Και να αναφέρουμε τις προσδοκίες μας σε σχέση με τις προτάσεις της Κομισιόν. Είναι επίγον το θέμα, γιατί αν δεν αλλάξει τίποτα, η Κομισιόν τον Νοέμβριο περίπου θα παρουσιάσει την πέμπτη της περιφερειακή έκθεση, στην οποία θα παρουσιαστεί και η πολιτική συνοχή μετά το 2013. Αν θέλουμε λοιπόν να μπορέσουμε να επιδράσουμε επί των εξελίξεων, θα πρέπει κάτι να κάνουμε μέσα στη συνεδρία της Επιτροπής μας και μέσα στα πλαίσια των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας. Να έχουμε τώρα αυτό το ανεπίσημο έγγραφο, όπως σας είπα, και μετά το καλοκαίρι να συγχειρήσουμε μέσα στα πλαίσια της ομάδας εργασίας, να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και να έχουμε τελικά κάποια πρόταση που θα αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες μας και τις προσδοκίες μας. Uh, um, Αυτά για την ενημέρωσή σας. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις και σχόλια, θα ήθελα να σας πω ότι αύριο θα αρχίσουμε να συνεδριάζουμε στις 9 και θα πρέπει να έχετε τις κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί έχουμε την έκθεση ε, ε, να ψηφίσουμε. Κυρίλοφ και Γιάνν Όλμπριχ. Τώρα έχουμε συνεδρία συντονιστών για μισή ώρα. Παρακαλώ τους να περιμένουν στην αίθουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. No, esto, no sé si lo ha dicho Adrede o es que da igual, no pasa nada porque lo haremos.